βρεθεί ανάμεσά μας και οι υπόλοιποι αντιπρόεδροι απουσίαζαν, ε, απουσιάζουν μάλλον και γι' αυτό προεδρεύω εγώ σήμερα το πρωί της συνεδρίασης. Ναι, εκτιμώ ιδιαίτερα το ότι βρίσκεστε εδώ, αλλά θα ήθελα να διαμαρτυρηθώ έντονα επειδή ανεβλήθη η συνεδρίαση των συντονιστών λόγω της απουσίας της Προέδρου. Θα πρέπει να διατηρούμε το πρόγραμμά μας και τον προγραμματισμό της συνεδρίασης. Αυτό θα πρέπει να γραφτεί και στα πρακτικά και να πούμε ότι είναι απαράδεκτο την προηγούμενη μέρα ή μάλλον και μία εβδομάδα ακόμα πριν δεν ε, θα έπρεπε να ακυρώνονται αυτές οι συναντήσεις επειδή η Πρόεδρος ε, δεν μπορεί να παραβρεθεί. Λυπάμαι, είμαι πολύ, μα πολύ θυμωμένη. εντάξει θα διαβιβάσουμε την δήλωσή σας, αλλά όπως βλέπετε αυτά συμβαίνουν ανεξαρτήτως από την βούλησή μου. Εν υπάρχουν κάποια σημεία που πρέπει να έχουμε υπόψη μας στην σημερινή μας συνεδρία. Θα ξεκινήσουμε τις εργασίες ε, με την παρουσίαση του κυρίου Διαμαντούρου, του Ευρωπαίου Διαμασολαβητή, για την ε, έκθεση δραστηριοτήτων ε, του η ε, κυρία Ντεσέβα ε, έχει οριστεί ως τη συγγήτρια και θα φτάσει από λεπτό σε λεπτό. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν ε, καθυστερήσαμε και επειδή έχουν γίνει κάποιες αλλαγές στη μεσαδιάταξη, γι' αυτό και έχει καθυστερήσει. Μετά θα έχουμε την παρουσίαση των κύριων Διαμαντούρ της ειδικής έκθεσης για την οποία έχει διοριστεί ως η κυρία Παλιαδέλη. Τα σημεία 6, 7 και 8 αναβάλλονται. Το σημείο 9 που αφορά την αποστολή στην Καμπανία θα εξεταστεί σήμερα το απόγευμα γύρω στις 16.00 ε, μετά από το σημείο 14. Το σημείο 12 θα μας το περιουσιάσει ο αναφέρον κύριο Στόκουελ. Θα πρέπει να πούμε ότι στο παρελθόν το Κοινοβούλιο ήδη υποστήριξε τους ε, ε, αναφέροντες για τον Λόιντ μετά από έκθεση του κύριου Πέρι και ο ε, φάκελος αυτός αρχιοθετήθηκε, αλλά εν υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα σχετικά με την εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου από πλευρά ε, ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και από πλευρά του κράτους μέλους και γι' αυτό ο κύριος Στόκελ υπέβαλε αυτή την αναφορά. Το σημείο 13 θα το εισαγάγει η κυρία Γκέριγκερ και σήμερα το απόγευμα μετά από τις συνεδρία των συντονιστών Παρατήρησε εκτός μικροφώνου. Ε, κατάλαβα καλά, το υπόθεση Λόιτ θα μεταφερθεί και αυτή στο απόγευμα. την συνεδρίαση. Όχι, όχι, μα σήμερα το πρωί, σήμερα το πρωί θα εξεταστεί ε, η υπόθεση αυτή. Λοιπόν, σήμερα το απόγευμα μετά τη συνεδρίαση των συντονιστών που θα διεξαχθεί μεταξύ 2.30 και 3 το μεσημέρι θα έχουμε την παρουσίαση των μελετών σχετικά με την επιστροφή περιουσιών μετά από αναφορές ε, πολλών ε, αναφερομένων πολλών αναφερόντων οι οποίοι θα είναι παρόντες, επαναλαμβάνω, και θα λάβουν το λόγο κατά τη διάρκεια της ε, συνεδρίασης. Ο κύριος παραδιάστα θα είναι παρόν ε, και ο κύριος ε, Περμέγερ. Λοιπόν, με αυτές τις αλλαγές προτείνω να υιοθετήσουμε τη μερίστα διάταξη. Ευδευλημένο είναι αυτό το που σας ζητώ, εντάξει. παρατήρηση εκτός μικροφώνου. Η Πρόεδρος ε, κάνουμε ό,τι μπορούμε σήμερα το πρωί. Και θα περάσουμε τώρα στην παρουσίαση του κύριου Διαμαντούρου. Σας ευχαριστούμε για την ε, παρουσία σας και θα ακούσουμε την ε, ετήσια έκθεση σας για το 2009. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρα. Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος που είμαι σήμερα και που εργαζόμαστε υπό την Προεδρία σας. Πρόεδρε, <clears throat> αξιότιμα μέλη, Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μου δίνετε να σας μιλήσω για την ετήσια έκθεσή μου ε, το έτος 2009. Ε, Υπάρχουν στατιστικά βασικά νούμερα, βασικά στοιχεία από προσφυγές προσώπων μη κυβερνητικών οργανώσεων, ενώσεων ε, το 2009. Υπέβαλα στον πρόεδρο Μπούζεκ την έκθεση 19 Απριλίου. Η έκθεση αυτή βεβαίως είναι η πρώτη ετήσια έκθεση που έχω την τιμή να σας υποβάλω αφότου με τίμησε με το Κοινοβούλιο επανεκλέγοντας με τον Ιανουάριο πάλι στη θέση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή. Ε, είμαι ευγνώμων για την εμπιστοσύνη του Κοινοβουλίου και σας διασφαλίζω, σας διαβεβαιώνω ότι θα συνεχίσω να συνεργάζομαι στενά με την Επιτροπή για τον κοινό στόχο της προσφοράς στους Ευρωπαίους πολίτες των μέγιστων ωφελών στα πλαίσια των συνθήκων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ διερευνώ ε, προσφυγές κακοδιοίκησης που ε, είναι ένας ευρύτατος ε, τομέας ε, από καθυστερημένες πληρωμές έργων της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την άρνη, μέχρι την άρνηση χορήγησης εγγράφου ή πληροφορίας ή μη απάντηση σε μια επιστολή. Αντίθετα με τις αποφάσεις του δικαστηρίου δεν είναι νομικά δεσμευτικές οι αποφάσεις μου, όμως με την πειθό προσπαθώ να εξεύρω φιλικαίους διακανονισμούς και λύσεις που θα καλύπτουν τα δύο μέρη. Οι υπηρεσίε μου έτσι είναι πιο ευέλικτες και ταχύτερες καμιά φορά από ό,τι των δικαστηρίων. Και ένα πολύ σημαντικό για πολλούς προσφεύγοντες, οι υπηρεσίε που παρέχω είναι δωρεάν. Μετά την παρέμβασή μου τα θεσμικά όργανα ε, διακανονίζουν ε, τις διαφορές, και θέτουν τέλος σε ε, διακρίσεις. Ε, πήρα ε, πολλές επιστολές 3.098 από διάφορες πηγές και αυτό είναι το 10%, 10 λιγότερες προσφυγές σε σχέση με το 2008. Ίσως εκπλαγείτε ακούγοντας ότι αυτό αυτή η μείωση είναι ενθαρρυντική και θα εξηγήσω σε λίγο γιατί. Προσπαθώ να βοηθώ κάθε προσφεύγοντα στο διαμεσολαβητή ακόμα και αν δεν είναι η προσφυγή στα πλαίσια της εντολής μου. Τον Ιανουάριο του 2009 άρχισα, έβαλα στην ιστοσελίδα μου έναν οδηγό ε, διαδραστικό και στις 23 γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο οδηγός ε, δίνει οδηγίες στον προσφεύγοντα για να απευθυνθούν στον κατάλληλο φορέα ή αρχή, είτε σε μένα ή στον ε, ε, εθνικό συνήγορο ή στο, μέσα από το δίκτυο Solved. Από την έναρξή του στις 5 Ιανουαρίου και μέχρι το τέλος του 2009 ο οδηγός έδωσε συμβουλές σε πάνω από 26.000 χρήστες. Τώρα το νούμερο είναι 33.000 πλέον. Σε αυτή την περίοδο 1.413 χρήστες του οδηγού ε, πήραν τη συμβουλή να απευθυνθούν στην Επιτροπή Αναφορών. Αυτή ήταν η συνηθέστερη συμβουλή. Η μείωση του συνολικού αριθμού των ε, προσφυγών δείχνει ότι ε, επικουρούμενοι από τον οδηγό, πιο πολλοί πολίτες βρίσκουν τη σωστή ε, διεύθυνση για να απευθυνθούν την πρώτη φορά, έτσι μειώνουν τον αριθμό των μη παραδεκτών αναφορών, που ήταν ένα παλιό αίτημα του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής σας προς τον Διαμεσολαβήτη. Μην υποτιμούμε πόσο σημαντικό είναι να κατευθύνονται στην αρμόδια αρχή ευθύ εξ αρχή οι πολίτες και να μην έχουν τι απογοητεύσει τι καθυστερήσει, ε, όταν διαπιστώνουν ότι κατέθεσαν την ε, προσφυγή σε λάθος φορέα. Έτσι οι προσφυγές επιλύονται αποτελεσματικά και μπορούν να έχουν τα και να τα ασκούν επίσης μειώνοντας το ποσοστό των μη παραδεκτών αναφορών η δική μου αρχή βοηθάει καλύτερα τους προσφεύγοντες με παραδεκτές αναφορές. Τα αποτελέσματα του γραφείου μου για αυτά τα ε, πρόσωπα ε, είναι ό,τι καλύτερο έχει επιδείξει το έργο μου. Πιστεύω ότι με το διαδραστικό οδηγό οι πολίτες ε, δέχονται βελτιωμένες υπηρεσίες από εμάς. Το 2009 το γραφείο μου έκλεισε 318 ε, έρευνες, οι περισσότερες, το 70% δηλαδή ολοκληρώθηκε μέσα σε ένα χρόνο. Πάνω από το μισό 55% ε, τελείωσαν μέσα σε τρεις μήνες. Κατά μέσον όρο οι έρευνες ε, πήραν για να ολοκληρωθούν εννέα μήνες. Οι περισσότερες έρευνες αφορούσαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μετά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το Ευρωπαϊκό Γραφείο Επιλογής Προσωπικού και το Συμβούλιο. Ε, με ικανοποίηση σημειώνω ότι το 2001 το 56% όλων των ερευνών ε, ε, έκλεισαν είτε από το, τη δική μου αρχή ή ε, επιλήθηκαν φιλικά. Αυτό είναι μεγάλη βελτίωση σε σχέση με το 2008 όπου το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 36% σε 35 περιπτώσεις έκανα κάποιες κριτικές παρατηρήσεις. Και αυτό και είναι μεγάλη πρόοδος σε σχέση με το 2008 όπου έκανα κριτικές παρατηρήσεις σε 44 υποθέσεις και το 2007 όπου 55 τέτοιες ε, παρατηρήσεις εκδόθηκαν. Η συνεχιζόμενη μείωση είναι καλό νέο, όμως ακόμα είναι πολλές. Σε ό,τι αφορά την προέλευση των αναφορών θα δείτε λεπτομέρειες ε, αναχώρα στην ετήσια έκθεση και στο χάρτη και τα στοιχεία που έχει η τελευταία σελίδα της ανασκόπησης που ελπίζω να έχετε στη γλώσσα σας. Όταν ένα θεσμικό όργανο δεν ανταποκρίνεται στις, στις προτροπές μου σε θέματα θεμελιώδων αρχών, Τότε ε, παραπέμπω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2008 έστειλα μια τέτοια έκθεση στο Κοινοβούλιο σχετικά με διακρίσεις λόγω ηλικίας στην Κομισιόν. Και με ικανοποίηση παρατήρησα ότι αυτή η Επιτροπή ασχολήθηκε ε, άμεσα με την ε, αναφορά αυτή, την έκθεση αυτή και η έκθεση Μεντίνα που, Ματίνα που εγκρίθηκε από την Ολομέλεια ε, με κάλυψε τελείως. Τα τελευταία χρόνια έκανα μεγάλες προσπάθειες για να ε, βελτιώσω τις υπηρεσίες προς επιχειρήσεις, μη κυβερνητικές οργανώσεις, ενώσεις, ε, περιφερειακές αρχές και άλλες ομάδες στόχο. Δηλαδή προς οποιονδήποτε που ενέχεται σε προγράμματα ή έργα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει άμεση συνεργασία με ενωσιακές αρχές. Το 2009 προσπαθήσαμε ακόμη περισσότερο περισσότερο για να καλύψουμε κι άλλους προσφεύγοντες και να οργανώσουμε σειρά εκδηλώσεων με μη κυβερνητικές οργανώσεις, ε, επιχειρηματικές ε, μονάδες, ε, ομάδες συμφερόντων κλπ. Ε, έχουμε 85% αύξηση της κάλυψης από τα μέσα του έργου του διαμεσολαβητή το 2009. η αύξηση των, του αριθμού των ερευνών από 293 σε 335 στηρίζεται σε προσφυγές από το 2009, αλλά εν μέρει αποδίδεται και σε αυτές τις δραστηριότητες. Για να ε, κοινοποιηθεί καλύτερα το έργο του διαμεσολαβητή, κατά τη διάρκεια του έτους συνεργαστήκαμε και με άλλα δίκτυα επίλυσης διαφορών και πληροφορικά δίκτυα, όπως το Solve, το Europe Direct. Το 2009 ε, το πιο σύνηθες πρόβλημα ήταν η έλλειψη διαφάνειας στην ε, διοίκηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό υπήρχε στο 36% στις ε, έρευνες και υπήρχε και συμπεριλάμβανε και άρνηση παροχής εγγράφων. Άλλα θέματα κακοδιοίκησης, κακοδιαχείριση ήταν καθεστημένες πληρωμές, κατάχρηση εξουσίας, προβλήματα διαδικαστικά κλπ. Ε, ένα παράδειγμα από αυτή την τελευταία κατηγορία. Επέκρινα την Κομισιόν γιατί δεν έκανε σωστή σημείωση ε, με, από μια συνάντηση στον ΤΕΛ με έναν ε, κατασκευαστή κομπιούτερ. το υπήρχε θέμα με τον ανταγωνιστή και είπα ότι η Κομισιόν θα μπορέσει να βελτιώσει τη διαχείριση και οι έρευνες αντιτράστα θα έπρεπε να τεκμηριώνονται στο μέλλον πλήρως. Με κάποια ανησυχία σημείωσα στην έκθεσή μου το υψηλό ε, ποσοστό προσφυγών λόγω της έλλειψης διαφάνειας. Ε, μια υπόλογη διαφανής ε, διαχείριση είναι απαραίτητη για να έχει την εμπιστοσύνη των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από την πλευρά μου θα συνεχίσω να επιμένω στο θεμελιώδες δικαίωμα πρόσβαση στα έγγραφα που προβλέπεται στο άρθρο 42 του χάρτη, το άρθρο 15 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και Διαβεβαιώνω ότι το δικαίωμα πρόσβαση στον διαμεσολαβητή και τη υποβολή αναφορά στο Κοινοβούλιο με βάση τα άρθρα 43 και 44 του χάρτη είναι, πρέπει να είναι γνωστά και να αξιοποιούνται ούτω ώστε να προσφεύγουν και να ζητούν αποζημίωση. Η συνθήκη της Λισαβόνας τώρα προβλέπει νέα ε, συμμετοχή δημόσια. Πρόκειται για την ε, πρωτοβουλία των πολιτών. Είμαι πεπισμένος ότι αυτό θα συμβάλλει σημαντικά στην ενίσχυση των Ευρωπαίων πολιτών. Στις αρχές του χρόνου απάντησα στη δημόσια διαβούλευση προβάλλοντας συγκεκριμένες προτάσει για την πρωτοβουλία των πολιτών και πώς θα πρέπει να λειτουργεί στην πράξη. Είναι σημαντικό να προβλέψουμε τυχόν ε, προβλήματα και ερωτηματικά, ιδιαίτερα αυτά που μπορούν να ε, οδηγήσουν σε προσφυγή στο διαμεσολαβητή, εντοπίζοντας τέτοια ερωτήματα εκ των προτέρων, προτείνοντας αποτελεσματικές λύσεις, λύσεις θέλω, στοχεύω στην καλή διοίκηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την πλήρη αξιοποίηση του πολύτιμου εργαλείου για τους πολίτες. Επίση, επίσης, στόχος μου είναι να διασφαλίσω ότι οι εκπρόσωποι των πολιτών, η κοινωνία των πολιτών θα ωφεληθούν από τις νέες διατάξεις της συνθήκης σχετικά με τις διαβουλεύσεις, το διάλογο και την δυνατότητα κοινοποίηση και δημόσιας ε, ενημέρωσης σχετικά με τις απόψεις τους. Επίσης, σημειώνω ότι η συζήτηση σχετικά με του κανόνε πρόσβαση στα έγγραφα είναι πολύ σημαντικό θέμα για την διαφάνεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν δεν παρακολουθήσατε τη συζήτηση σας θυμίζω ότι η Κομισιόν πρότεινε μέχρι τώρα αλλαγέ στην τωρινή πρόσβαση στα έγγραφα που πιστεύω ότι θα οδηγήσει σε πρόσβαση σε λιγότερα και όχι περισσότερα έγγραφα. Το Μάρτιο του 2009 το Κοινοβούλιο ενέκρινε την έκθεση Κάσμαν που ε, ε, κάλυψε πολλά προβλήματα που είχα και εγώ και ζήτησε από την Κομισιόν να τροποποιήσει τις προτάσεις της. Ελπίζω ότι η πρόταση της Κομισιόν θα τροποποιηθεί όντως ούτως ώστε να υπάρχει η ευρύτερη δυνατή πρόσβαση στα έγγραφα από τους πολίτες και άλλους εμπλεκομένους. Ένα άλλο ανησυχητικό θέμα αφορά προβλήματα που έχει η Κομισιόν στην έγκαιρη πληρωμή των λογαριασμών της σε τρίτους όπως αναδόχους τα τελευταία χρόνια έλαβα πάνω από 30 προσφυγές για καθυστερημένες πληρωμές από κυβερνητικές οργανώσεις, ερευνητικά κέντρα, εταιρείε, ενώσεις και άλλες οργανώσεις. Το 2008 διεξήγαγα έρευνα για αυτό το θέμα που επιβεβαίωσε ότι αν και επετελέστη πρόοδο τα τελευταία χρόνια, οι καθυστερούμενες πληρωμές εξακολουθούν να συνιστούν σοβαρό πρόβλημα στην Κομισιόν. Και μάλιστα έγιναν καθυστερήσεις σε μία περίπτωση από 5, δηλαδή στο 20% όλων των περιπτώσεων το Μάρτιο του 2009 άνοιξα λοιπόν μία έρευνα ε, συνέχισης follow-up για να δω Ποια μέτρα έλαβε η Κομισιόν πρόσφατα για να αντιμετωπίσει το θέμα των καθυστερούμενων πληρωμών. Και με ικανοποίηση σημειώνω ότι τον Απρίλιο του 2009 άρχισε νέα πρωτοβουλία από την Κομισιόν για, με στόχο τις ταχύτερες πληρωμές ε, για συμβάσεις. Ε, περαιτέρω βελτιώσεις θα πρέπει να λάβουν χώρα το ταχύτερο δυνατό, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά πιο ευπαθείς αν θέλετε αναδόχους όπως μεμονωμένα πρόσωπα, μικρομεσαίες επιχειρήσεις ή μη κυβερνητικέ οργανώσεις το Δεκέμβριο του 2009 ως μέρος της συμβολής μας για τη δημόσια διαβούλευση για το δημοσιονομικό κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπογράμμισα ότι οι σχετικοί κανόνες πρέπει να λαμβάνουν υπόψη το άρθρο 41 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων δίνοντας συμβουλές και καθοδήγηση στους, ε, ε, στους υπαλλήλους για το πώς θα έχουν υγεία δημοσιονομική διαχείριση και καλή διαχείριση. Ε, παράδειγμα, ο δημοσιονομικός κανονισμός θα πρέπει σε εξαιρετικές περιπτώσεις ε, να προβλέπει εξκρέσια ε, πληρωμές ε, ως αποζημίωση για σοβαρά προβλήματα τα οποία προκάλεσε η κακοδιοίκηση. Η μεταρρύθμιση του δημοσιονομικού κανονισμού είναι εξαιρετική ευκαιρία ούτως ώστε να το θεμελιώδες δικαίωμα για την καλή διακυβέρνηση να τεθεί σε εφαρμογή. Θέλω να εξηγήσω τώρα τι επιτυγχάνουμε σε ό,τι αφορά τους στρατηγικούς στόχους που ανέφερα σε προηγούμενες παρουσιάσεις μου σε αυτή την Επιτροπή από τότε που ανέλαβα τα καθήκοντά μου το 2003 ανέπτυξα και αναδιάρθρωσα το γραφείο για να υπηρετώ τους πολίτες των 27 κρατών μελών σε 23 ε, επίσημες γλώσσες. Θα πρέπει επίσης οι πολίτες των υποψηφίων χωρών να παίρνουν στην γλώσσα τους τις πληροφορίες που ζητούν. Είμαι προφανώς ευγνώμων για την υποστήριξη την οποία το Κοινοβούλιο ως ε, αρχή δημοσιονομική ε, μου προσέφερε αντιδρώντας θετικά στα αιτήματα επί του προϋπολογισμού που διατύπωσα για να έχω υψηλή ποιότητας υπηρεσίες σε συνεχιζόμενη πολυετή βάση προγραμματισμού συνέχισα τις προσπάθειές μου για να βελτιώσω την ποιότητα των πληροφοριών προς τους πολίτες και τους πιθανούς προσφεύγοντες σε βάση του, του ενωσιακού δικαίου. Πολύ από αυτό το έργο έγινε από το δίκτυο του διαμεσολαβητή που περιλαμβάνει και αυτή την επιτροπή και αποτελείται από 94 γραφεία σε 32 χώρες που καλύπτουν ε, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το εθνικό επίπεδο στις χώρες που έχουν υποβάλει αίτηση ε, και την Νορβηγία, την Ισλανδία και πρόσφατα και την Ελβετία. Συνεργάζεται σε ημερήσια βάση για την διευθέτηση των υποθέσεων και σε συνεχιζόμενη βάση ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μέσα από σεμινάρια, εκδηλώσεις, newsletters, ε, ενημέρωση, ηλεκτρονικό φόρουμ συζητήσεων και ηλεκτρονική υπηρεσία ειδήσεων. Ένα στόχο του δικτύου είναι να διευκολύνει την ταχεία μεταφορά των προσφυγών στον, στον αρμόδιο ε, ε, συνήγορο. Η κοινοτική διάσταση των διαμεσολαβητών θα πρέπει να ε, γίνει ευρύτερα γνωστή και να βελτιωθούν οι υπηρεσίε που παρέχονται στους προσφεύγοντες στα πλαίσια του, του ενωσιακού δικαίου. Υπάρχει μια δήλωση του Οκτωβρίου η οποία ε, υπάρχει σε 23 γλώσσες από την ιστοσελίδα του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή. Το, υπάρχουν πολλά σεμινάρια που έχουν το, το σεμινάριο του Απριλίου στην Κύπρο το 2009 μας έδωσε μια ακόμα ευκαιρία να βελτιώσουμε τη συνεργασία μας. Κυρία Πρόεδρε, ε, συνεχίζω να προσπαθώ για να διαβεβαιώσω ότι οι ευρωπαϊκοί φορείς θα έχουν μια προσέγγιση σε, όλες, ε, σε όλους τους τομείς βασισμένη προς τον πολίτη, ε, επιδιώκοντας πάντα φιλικές λύσεις και ε, κάνοντας περισσότερες έρευνες ε, με δική μου πρωτοβουλία για να εντοπίσω προβλήματα και να ενθαρρύνω τις βέλτιστες πρακτικές. Για να προωθήσω το στόχο αυτό σε σχέση με την Κομισιόν συνεχίζω να αναπτύσσω τις ε, επαφές μου με τους αρμόδιους επιτρόπους και έκανα συναντήσεις με τους γενικούς διευθυντές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπως και με το Γενικό Γραμματέα. Το 2009 ενέκρινα μία δήλωση αποστολής για τον φορέα μου, η οποία έχει ως εξή και παραθέτω. Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής επιδιώκει δίκαια αποτελέσματα μετά από προσφυγές κατά των κοινωτικών θεσμικών οργάνων και τάσεται υπέρ της διαφάνειας ε, στην κουλτούρα της υπηρεσίας του. Θέλει να δημιουργηθεί εμπιστοσύνη μέσα από το διάλογο μεταξύ των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να προαγάγει τα υψηλά ε, πρότυπα ε, συμπεριφοράς στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά το τρέχον έτος προτίθεμαι να καταρτήσω έγγραφο στρατηγική το οποίο θα αναφέρει τις αρχές που αναφέρει το, η δήλωση αποστολής και θα καλύψει την πενταετή εντολή του διαμεσολαβητή. Παρ' όλα αυτά, ο διαμεσολαβητής δεν μπορεί να εργάζεται μόνος ε, για να η διασφάλιση ε, βέλτιστης διαχείρισης ε, θα πρέπει να επιτευχθεί μαζί με τα, μέσα από συνεργασία με τα θεσμικά όργανα. Θα πρέπει να μαθαίνουμε από λάθη, να έχουμε σωστούς μηχανισμούς, θα πρέπει να εργαζόμεθα με διαφάνεια. Αυτά είναι τα πολύ σημαντικά μέσα, ούτως ώστε να οικοδομηθεί εμπιστοσύνη μεταξύ πολιτών. Οι περισσότερες ε, υποθέσεις που επιλύθηκαν φιλικά είναι πηγή μεγάλης ενθάρρυνσης για μένα ακριβώ επειδή συνιστούν απτή απόδειξη αυτής της συνεργασίας μεταξύ των θεσμικών οργάνων και του διαμεσολαβητή. Κυρία Πρόεδρε, με τη δική σας ε, υποστήριξη και την υποστήριξη και την καθοδήγηση της Επιτροπής ε, θα ε, στηριχθώ στα επιτεύγματα του παρελθόντος έτους ούτως ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να έρθει πλησιέστερα στους πολίτες και να αποκτήσει ανθρώπινο πρόσωπο η ενωσιακή διοίκηση. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε κύριε Διαμαντούρο για την έκθεσή σας αλλά και για το σύνολο των εργασιών σας και πράγματι κατανοούμε ότι θέλετε να βρίσκεστε όσο πιο κοντά γίνεται στον Ευρωπαίο πολίτη, κάτι το οποίο προσπαθούμε να πετύχουμε και εμείς στην Επιτροπή Αναφορών. Σας ευχαριστούμε λοιπόν και για την συνεργασία σας εδώ και μερικούς μήνες ε, αλλά έχω παρατηρήσει ότι δίνεται ψυχή και σώμα σε αυτήν την εργασία που έχετε αναλάβει το, το έργο σας να δώσω το λόγο στην ε, Επιτροπή κυρία Κώστα Ρόζα από την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλή σας ημέρα ευχαριστώ κύριε Διαμαντούρο για την παρουσίαση της ετήσιας εκθέσεώς σας Μιλήσατε για τη σχέση σας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, άρα δεν μου αφήνετε και ιδιαίτερα περιθώρια να πω πολλά πράγματα, διότι συμφωνούμε με τα περισσότερα των όσων είπατε. Δράτω με τις ευκαιρίες, προκειμένου σας συγχαρώ για την επανεκλογή σας, αν και πραγματοποιήθηκε την 20η Ιουνίου, ε, Ιανουαρίου συγγνώμη, η ιουνιου έχει ξεκινήσει πολύ νωρίτερα, Ιούλιο-Αύγουστο του προηγούμενου έτους. Να τονίσω πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ο βασικός πελάτης του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή λόγω της φύσης των αρμοδιοτήτων του και εκφράζει την ικανοποίησή της πως φέτος, δηλαδή στην έκθεση του 2009, ο αριθμός των προσφυγών μειώθηκε κάτι το οποίο αποδεικνύει ότι και η Κομισιόν από πλευρά τη καταβάλει προσπάθειες ε, προκειμένου να ε, επιληθούν οι διαφορές φιλικά ή και να μπορεί να αποζημιώσει τον ε, προσφεύγοντα. Είμαστε λοιπόν στην υπηρεσία της κοινωνίας γενικότερα. Να πω επίσης σε ό,τι αφορά τα του οίκου μας ότι ο κύριος Γεμαντούρος ε, συνάντησε την κυρία Ντάι, η Γενική Γραμματέα της Επιτροπής, ε, πέρυσι και είχε την ευκαιρία να συναντήσει και τους γενικούς διευθυντές σε μια συνάντηση τον, που διεξήγησε τον Απρίλιο ή τον Μάιο, αν δεν σπάλλω, τη περασμένης χρονιά, που ήταν ιδιαίτερα επικοδομητική και στην οποία δώσαμε συνέχεια μετά από ανάληψη πρωτοβουλειών εντός ε, του οίκου μας ε, και όπως είπε ο κύριος Διαμαντούρος ε, συχνά συνέβαλε στο να μεταφέρει στους γενικούς διευθυντές ότι το έργο του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή είναι να ενισχύσει, να δημιουργήσει μια κουλτούρα υπηρεσιών, προσφοράς υπηρεσιών και όχι μια κουλτούρα παραπώνων και επίρρηψη ευθυνών. Ε, ακόμα και αν αναφερόμαστε στην έκθεση του 2009 θα ήθελα να παρατηρήσω ήδη πως ο κύριος Διαμαντούρος θα συναντήσει την, ε, το σώμα της Επιτροπής ε, φέτος αυτό δεν θα γίνει άμεσα διότι δεν έχει ολοκληρωθεί η σύνθεση των υπηρεσιών του κάθε επιτρόπου, δεν ξέρουμε ποιος κάνει τι ακριβώς. Η ατζέντα είναι ιδιαίτερα φορτωμένη, αλλά αυτή η συνάντηση, το ορκίζομαι, θα πραγματοποιηθεί φέτος. Και κάτι άλλο, να σας ευχαριστήσω για την ευελιξία σας σχετικά με την telephone procedure δηλαδή την επίλυση των ερευνών με τηλεφωνική συνδιάλεξη. Αυτό είναι κάτι το οποίο ε, έδειξε την αποτελεσματικότητά του, μπόρεσαν να επιληθούν τάχιστα κάποια θέματα που διαφορετικά θα χρονοτριβούσαν. Να σε ευχαριστήσω επίσης για το γεγονός ότι οι προσφυγές ε, εξετάζονται ακόμη πιο γρήγορα από το παρελθόν. Ε, υπάρχουν κάποιες διαδικασίες που βλέπουν την, συνεργασία, την διαβούλευση με την Κομισιόν και με τον αναφέροντα. Ε, σας ευχαριστώ επίσης για τις επαφές με το Solvit και τις συνεδριάσεις που είχατε με αυτούς και με το Europe Direct και την Γενική Διεύθυνση Εμπορίου. Να υπογραμμίσω επίσης μισό λεπτό γιατί το ξέχασα. Α, ναι, την εκστρατεία πληροφόρησης ε, που έχετε αναλάβει. Πραγματικά διαδώσατε το ζήτημα σε όλες ε, τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, ακόμα και στις ε, στους μελλοντικούς μελλοντικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσένταξη χώρες δεν θα ήθελα το να μακρηγορήσω όμως διότι πιστεύω πως ε, όλοι μας καταλάβαμε ότι η έκθεση αυτή ήταν ιδιαίτερα καλή και αποτελεσματική. Ο μεσολαβητής ε, διαφέρει με το δικαστήριο διότι μπορεί να αναλάβει κάποιες έρευνες ε, μετά από πρωτοβουλία του και έχει την εξουσία να έρευνα και να θέτει το δάχτυλο επί των τύπων των ύλων και να γνωρίζει τι ακριβώς συμβαίνει για να μπορέσουν τα πράγματα να έρθουν στη θέση τους, να επανέλθουν στη θέση Ευχαριστώ. Ε, σας ευχαριστώ για τις προφορίες ε, και όντως ε, μας αποδείξατε ότι έχετε μια πολύ καλή συνεργασία με τον διαμεσολαβητή μας. Μας ενδιαφέρει πολύ το θέμα διότι για έναν Ευρωπαίο πολίτη όταν τα κάτι δεν πάει καλά είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν πάει καλά. Πρέπει να αλλάξουμε λοιπόν αυτή την εικόνα. Χρειάζεται όλοι μαζί να προσφέρουν την καλύτερη δυνατή υπηρεσία προς τους πολίτες μας. Ευχαριστώ. Θέλετε να λάβετε λόγο κύριε Διαμαντούρο. Κύριε Πρόεδρε, είμαι στα χέρια σας. Εάν θέλετε να ακούσουμε πρώτα τους συναδέλφους σας, να σημειώσω τις παρατηρήσεις τους και εν συνεχεία να απαντήσω. Σημείωσα αυτά που είπε η κυρία Κωνσταρόζα και θα απαντήσω μετά από δύο-τρεις ακόμα παρεμβάσεις. Θα ξεκινήσω δίνω τον λόγο στην κυρία Νίντελ Σέβα που είναι η συγγήτριά μας και η ε, κυρία Μόκεν και ο κύριος Κάσμαν έχει στήσει το λόγο. Ίσως ε, να ακούσουμε τώρα τρεις ε, συναδέλφους και μετά να απαντήσετε. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κύριε Γεμαντούρο. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πρώτα τα όλα για την παρουσίαση, την εξαντλητική θα έλεγα, την αναλυτική που κάνετε και συμφωνώ απόλυτα με τα λόγια της Κομισιόν και θα ήθελα να σε ευχαριστήσω για την ετήσια έκθεσή σας του 2009. Να σε ευχαριστήσω επίση και για την εργασία σας εδώ στο πλαίσιο της Επιτροπής Αναφορών και τονίζω ότι η σημερινή σα παρουσία αλλά και η ε, παρακολούθηση των εργασιών τη Επιτροπή Αναφορών από πλευρά των υπηρεσιών σα δείχνει πόσο καλή είναι η συνεργασία ανάμεσα στα δύο θεσμικά όργανα, το Κοινοβούλιο και τον Διαμεσολαβητή. Και η συνεργασία αυτή είναι πολύ σημαντική το σου των μάλλον καθώ είναι και το σύμβολο, το σύμβολο του εισάμεση εκπροσώπηση των συμφερόντων και ενδιαφερόντων των πολιτών και όλα αυτά δεν τα λέω τυχαία διότι θα ήθελα να επενθυμίσω δύο πράγματα. Πρώτον, πως ε, και μέχρι τώρα δεν το είχα πράξει, να σας συγχαρώ για την <clears throat> επανεκλογή σας, το επενθυμίζω, διότι αναφέρομαι στην νομιμότητα του Κοινοβουλίου πάνω αυτά τα ζητήματα και που προσφέρει μια νομιμότητα ακόμα μεγαλύτερη στο πρόσωπό σα ε, Θα ήθελα να επενθυμίσω επίσης τη συνθήκη τη Λισαβόνα και τη νέα χάρτα των θεμελιωτών δικαιωμάτων και τον δεσμευτικό χαρακτήρα. Όπως είπατε πολύ σωστά στην έκθεσή σας, το αισθανόμαστε λοιπόν σαν μια κόκκινη γραμμή με την χάρτα των, των θεμελιωτών δικαιωμάτων. Έχουμε μια νέα πρόκληση ενώπιόν μα και οι εργασίε του Δημοσιολαβητή θα εκτιμηθούν έτσι περαιτέρω από του πολίτε και θα παρακολουθούν εκ του σύνεγγης από την Επιτροπή. Να ήθελα να υπενθυμίσω ότι συμφωνούμε απόλυτα με τις προτεραιότητές σας. Αυτές οι προτεραιότητες αποτελούν τμήμα των αξιών μας να, να προσπίσουμε τα θεμελιώδη δικαιώματα και να προωθήσουμε τη διαφάνεια και την πρόσβαση στα έγγραφα. Αυτό είναι κάτι το οποίο ακούγεται καθημερινά στις επαφές με τους πολίτες και σας ευχαριστώ για όλες τις προσπάθειες που καταβάλλετε προς την κατεύθυνση αυτή. Πράγματι, μας αναφέρατε τις ανησυχίες σας, μερικές δεν είναι καινούριε, αλλά ε, έφτασε η στιγμή να τονίσουμε την πρόοδο και τις επιτυχίες που έχουν γίνει και θα σας ενθαρρύνω να συνεχίσετε προκειμένου να καλύψετε τις λήψει τα κενά για να βελτιώσετε την λειτουργία και να επιφέρετε λύσεις που θα ικανοποιούν ακόμα περισσότερο τους πολίτες μας. Είτε πρόκειται για την μέση διάρκεια των ερευνών, δεν μπορώ παρά να την ικανοποίησή μου που η διάρκεια μειώθηκε και διαπιστώνουμε ότι έχει καταβληθεί ιδιαίτερη προσπάθεια. Είτε πρόκειται για την πρόσβαση στα έγγραφα ε, και τη δημιουργία της ε, ιστοσελίδας, ε, ότι αυτό πρέπει να τονιστεί. Επίσης, να σα συγχαρώ ε, σε ό,τι αφορά τις προκλήσεις, ε, άκουσα πολύ, πολύ ενδιαφέρον τις προκλήσεις που τονίσατε. Μιλήσατε για την ποιότητα της προφόρησης, την ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαμεσολαβητών, ε, ό,τι αφορά την Direct Europe και σίγουρα ο δημοσιολαβητής δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά του μόνος του. Εμείς είμαστε εδώ σε επιτροπή να σας πούμε ότι συμφωνούμε με αυτή την προσέγγιση που στηρίζεται στον πολίτη είναι, ε, συμβολίζει αυτή η ιδέα και το Ευρωκοινοβούλιο, αλλά όταν λέτε ότι το έργο του Δημοσιολαβητή είναι άρρηκτα συνδεμένο με τις σχέσεις του με τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα και ολοκρόνο λέγοντας πώς μπορείτε να βασιστείτε στην υποστήριξη της Επιτροπής Αναφορών και ελπίζω πως αυτή η συνεργασία που ήταν τόσο καρποφόρα μέχρι τώρα θα το συνεχίσει. Ευχαριστώ. Κυρία Όκεν. Δεν έχει ανοίξει το μικρόφωνο η κυρία Άουκεν. Είναι αναμένο, αναμένο είναι. Ήταν αναμένο, λέει κυρία Άουκεν, παρά το ότι δεν ήταν. Τέλος πάντων. Okay. Uh, and then not to repeat what just... Για να μην επαναλάβω το τα οποία προηγουμένω, απευθεία να σα δείξω κάποια προβλήματα θα πρέπει λοιπόν όλοι εδώ να πανηγυρίζουμε διότι άλλαξε γνώμη η Κομισιόν ε, ως ανάνητης υψίστης μια που έτσι έγινε. Τους αλλάξαμε γνώμη και αφού διαβάσαμε αυτή την τελευταία υπόθεση με μεγάλη μου χαρά ακούω ότι τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπε ότι συμφωνεί με τον διαμεσολαβητή. Οπότε, η διαφάνεια βεβαίως είναι ένα πάγιο πρόβλημα και θυμάμαι 20 χρόνια που ήμουν βουλευτήνα στο Δανέζικο Κοινοβούλιο παρά την σχετική νομοθεσία, παρά το ότι είχαμε διαφορετικές κυβερνήσεις από όλο το πολιτικό φάσμα, όλοι αυτοί λέγανε για το πόσο σημαντικό είναι και αυτό αφορά και τους ε, πολίτες όλους, όλους, όλους, διότι ε, κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να σταματήσουμε το πρόβλημα, το φαινόμενο αυτό, αλλάζαμε τους νόμους. Επομένως είναι για μια μάχη χωρίς τέλος. Ακόμα και όταν κανένας κερδίζει αυτή τη μάχη θα πρέπει να, είναι, να έχει με το όπλο παραπόδα. οπότε το ερώτημα είναι μπορούμε να κάνουμε τίποτε όσον αφορά το πρόβλημα. Πώς είναι στα αγγλικά? Letter of formal notice. Κάτσαν επιστολή όχλησης επίσημης. Και στη Δανία τώρα επομένως υπάρχει αυτό το πρόβλημα για το περιβάλλον. Οπότε θα πρέπει να ενεργήσουμε σύνομα σύμφωνα με την ε, παλαιότερη συνθήκη. Και η κόρη μου είναι στην ε, Επιτροπή και με το Περιβάλλον. Και μου είπανε, μαμά, όταν πας να δεις τον δημοσιολογητή, πες το. Γιατί αυτή η υπόθεση εκκρεμεί πολύ καιρό. Και οι πολίτες που έχουν εμπλακεί τελικά μείναν απ' έξω. Αυτό επομένως είναι πρόβλημα. Πρόβλημα επικοινωνίας. Καλά, και αν δεν μπορείτε να επαντήσετε τώρα, να τα πούμε κάποια άλλη στιγμή, αλλά παρακαλώ κάντε κάτι γι' αυτό επίσης. Μας είπατε και το θεωρώ πάρα πολύ θετικό. Το, το πώς γίνεται η συνεργασία με τα άλλα θεσμικά όργανα όπως την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και ξέρετε αυτή η τράπεζα δεν ε, δουλεύει μόνο στο εσωτερικό της Ένωσης αλλά και εκτός αυτής. Επομένως είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτή η αρχή να ε, συνεχίσει να ισχύει Και θα κάτσω και να διαβάσω το κείμενο γιατί μέχρι τώρα δεν είχα την ευκαιρία να το κάνω. Ευχαριστούμε. Κύριε Κάσμαν, έχετε το λόγο, λέει ο Πρόεδρο. Uh, uh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συγχαρητήρια κύριε Διαμαντούρο. Είναι πάρα πολύ αξιολόγη αυτή η έκθεση και πάρα πολύ σημαντικό το έργο που έχετε επιτελέσει. Συνήθω συμφωνώ με την κυρία Άουκεν, αλλά θα πρέπει να σα πω ότι για να αποδεχθεί κανεί ε, την έννοια του αμαρτήματος θα πρέπει κανένας να το αποδεχθεί και ιδεολογικά. Και εγώ είμαι άθεος. Παρόλα αυτά όμως, οπωσδήποτε, έχουν βελτιωθεί οι σχέσεις των θεσμικών οργάνων και οι σχέσεις μας με, τη, με τον Δημοσιολαβητή. Και τώρα, για να έρθουμε στο ψητό, έχουμε αυτό τον κανονισμό στον αφορά την προσβασιμότητα 1049 του 2001, που αφορά την προσβασιμότητα επομένως του κοινού στα επίσημα έγγραφα και όσον αφορά επομένως όλα αυτά που θέλουμε να δούμε και όπως σωστά μας είπατε υπάρχει εδώ μια επικάλυψη όσον αφορά τα περισσότερα αιτήματα προς εσάς ας πούμε για την επιλογή, τους διαγωνισμούς κλπ. Ερωτώ. Ποια θεσμικά όργανα τα περισσότερα έγγραφα, το Κοινοβούλιο, η Κομισιόν ή το Συμβούλιο η δε συνεργασία που έχετε με τα τρία όργανα πώς πάει. Επίσης, υπάρχει εδώ πέρα μια σύγκρουση μεταξύ προσβασιμότητα στα έγγραφα και από την άλλη μεριά προσβασιμότητα στις πληροφορίες. Και εδώ υπάρχει κάποια σύγκριση γιατί υπάρχει διαφορετική νομική βάση. Και δεν ξέρει ούτε ο κόσμος τι γίνεται ούτε με κυβερνητικές οργανώσεις. Και Εάν υπάρχει κάποιο θεσμικό όργανο το οποίο δεν ανταποκρίνεται στα αιτήματα τη προσβασιμότητα στα έγγραφα, θα πρέπει να επιληφθείτε και να εφαρμόσετε τον κανονισμό 1049 του 2001. Κύριε Διαμαντούρο, θα σας δώσω το λόγο και κατόπιν να ακούσουμε την κυρία Μπασέσκου και την κυρία ε, Ζντανόκα που έχει δει στο λόγο. Θέλετε τώρα να λάβετε το λόγο και να σας απαντήσει μετά και ο Διαμαντούρος. Καλά. Μπασέσκου. Mr. Diamandouros, I would like to congratulate you for the report that you presented us today. It's a pity though that most of... Ευχαριστούμε που ήρθατε εδώ να μας μιλήσετε και δυστυχώς εδώ πέρα λείπουν πάρα πολλοί συνάδελφοι και ο πρόεδρος ή η πρόεδρος της Επιτροπής μας. Επίσης θα πρέπει να σας πω και εγώ ίδια έχω καταλάβει ε, ότι πάρα πολύ σωστά λειτουργεί το, η υπηρεσία σας και την, τον περασμένο μήνα είχα καταθέσει κάποια αναφορά, κάποια καταγγελία, παράπονο και ευθύ αμέσω μου απαντήσατε και με ξεκάθαρο τρόπο. Μόνο ξέρω ότι δουλεύει η υπηρεσία σα όπω πρέπει. Όπω είπατε σωστά, η πρωτοβουλία των πολιτών είναι το να ξεκινήσει με καινούργια μορφή τη συμμετοχή δημοκρατία στην ΕΕ, ούτω ώστε υπάρχει μια εμπλοκή των πολιτών. Αλλά για πετε μα, κατά τη γνώμη σα, ποια είναι τα σημαντικότερα προβλήματα τα οποία θα προκύψουν εάν έχουμε τέτοιου είδου μέσα τέτοιου είδους πολιτική για τους πολίτες. Αυτό ήθελα συγκεκριμένα να σας ρωτήσω. Κυρία Κύριε Μπασέσκου, συμπαθάτε με, αλλά δεν κατάλαβα. ποιο, ποιο, ποιο μέσο πολιτικής, ποια πολιτική, για ποιο πράγμα αναφέρεστε. Η πρωτοβουλία των πολιτών, λέει η κυρία Μπασέσκου. Yes, Σας ευχαριστώ και εγώ θέλω να συγχαρώ τον κύριο Διαμαντούρο για την έκθεσή του. Um, uh, Μία πρόταση για ένα νέο νομοθέτημα. Έχουμε το άρθρο 298 τις συνθήκες που ορίζει για κάποια πρότυπα, κάποια στάνταρ υψηλά για το Μαθήση Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά εσείς τι λέτε. Με όλες αυτές τις κοινωνικές επιτροπές προσπαθούμε να ε, θεσπίσουμε ένα νέο κανονισμό όσον αφορά το προσωπικό τη υπαλλήλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καταλάβατε τι ρωτάω. Σε τι αναφέρεστε, λέει ο κ. Διαμαντούρο, αναφέρεστε στην, ε, στη θέσπιση, στη δημιουργία καινούριου διοικητικού δικαίου. Ναι, ναι, ναι, λέει η, κ. Δανόκα. Α, μάλιστα, κατάλαβα και θα σα απαντήσω. Και εννοώ, λέει η κ. Δανόκα, δεσμευτικά, νομικό, νομικά δεσμευτικό κανονισμό. Ευχαριστώ, λέει πρόεδρο, και τώρα να δώσουμε το λόγο. Ε, αν δεν σα πειράζει, κ. Διαμαντούρο σε, στον κύριο Ράφνερ που ζήτησε το λόγο. Yes, thank you. Only if you... Ευχαριστώ. Όχι, όχι, όχι, μπας και θέλετε να απαντήσετε πριν νωρίτες. Ό,τι θέλετε. Στη διάθεσή σας, λέει ο κ. Διαμαντούρος. Θα ήθελα να επανέλθω σε δύο σημεία στα οποία αναφερθήκατε όταν περίπου είχατε ολοκληρώσει την εισήγησή σας. Είναι δύο σημεία τα οποία σχετίζονται με ζητήματα που συζητήσαμε εδώ στο Κοινοβούλιο πρόσφατα, δηλαδή την τα στα έγγραφα. Το συζητήσαμε στην Επιτροπή Θεσμικών Θεμάτων και συντάσσουμε μια νέα έκθεση. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται για τεμάκι, κάπως έτσι ο συνάδελφος. Έτσι, ναι, ναι, ναι, ναι, έτσι. Και είχαμε και τον κύριο Κάσμαν που ασχολήθηκε Γι' αυτό σας λέω θα ήταν πάρα πολύ θετικό εάν ενσωματώναμε αυτά που μας είπατε εσείς εδώ και όλα όσα έχετε πει στο παρελθόν. Όλα αυτά να τα εντάξουμε στην έκθεση. Οπότε βοηθήστε μας παρακαλούμε να συντάξουμε την έκθεση αυτή. Με την πείρα σας. η πόρτα και, άρα, ή η υπόθεση πόρτα και άλλες υποθέσεις, ούτως ώστε να μπορούμε να έχουμε όσο γίνεται καλύτερη έκθεση. Γιατί πιστεύω ότι υπάρχει αυτή τάση που είπατε κι εσείς. Πόρσε, πόρσε ήταν αυτή η υπόθεση. Ε, γιατί έχουμε και τη δεδομένη στάση της Κομισιόν που δεν είναι και τέλεια. Πάρα πολύ θετικά ήταν τα όσα μας είπατε σχέση με, το, με την Πρασινή Βίβλα. Έχουμε τώρα το σχέδιο σχετικού κανονισμού. Οπότε θα σας καλέσουμε όταν έρθει η ώρα να έρθετε στην Επιτροπή μας και να μας τα πείτε. Επίσης, για πέστε μας, πώς βλέπετε το δικό σας ρόλο ως Ευρωπαϊκό Μεσολεύτη σε αυτή τη διαδικασία της Πρωτοβουλίες των πολιτών. Πρώτα-πρώτα όσον αφορά την αρχή της πρωτοβουλίας, όσον αφορά το παραδεκτό επίσης, γιατί στο σχέδιο κανονισμού η Επιτροπή λέει ότι κάποιες πρωτοβουλίες που στρέφονται κατά της Επιτροπής δεν θα πρέπει να επιτρέπονται. οι ανόητες, οι αβάσιμες πρωτοβουλίες. Το είπε και ο Επίτροπος Σεύκοβιτς. Όμως πώς θα κρίνεται από το παραδεκτό. Μήπως θα πρέπει ο διοσμελευτής να παίξει κάποιο ρόλο σε αυτό. Και επίσης, για κάποια πρωτοβουλία που ας πούμε έχει μαζέψει ένα εκατομμύριο υπογραφές και παρόλα αυτά η Κομισιόν την θεωρεί απαράδεκτη. Οπότε θα πρέπει να διαβαστεί η πρόταση στον Δημοσιολαβητή για να δούμε τι άλλου είδου γνώμη μπορεί να υπάρξει. Γιατί φοβάμαι ότι εάν ένα εκατομμύριο Ευρωπαίοι από όλη την Ευρώπη έχουν προσυπογράψει ένα κείμενο και καταλήγει να μην γίνεται τίποτα, αυτό είναι πρόβλημα. Πέστε μας παρακαλώ τις απόψεις σας. Ευχαριστώ πολύ. Θα ξεκινήσω μιλώντας στην Καλικίνο προκειμένου να απαντήσω στις ερωτήσεις που ετέθησαν ε, στην στα γαλλικά και μετά θα συνεχίσω στην αγγλική με τη σειρά λοιπόν που έλαβα τις ε, ερωτήσεις ε, θα προβώ και τις απαντήσεις. Ξεκινώντας λοιπόν να ευχαριστώ την κυρία Κώστα Ρόζα για τα καλά της λόγια. Χαίρομαι που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατανοεί και δέχεται τις ε, προσπάθειες που καταβάλει ο μεσολαβητής, ο διαμεσολαβητής ε, και που προσπαθούν να καταργήσει την ε, κουλτούρα των, της επιρρήψεως ευθυνών και των μομφών. Έλαβα λοιπόν τελευταία πολλά ενθαρρυντικά σχόλια για αυτό το έργο. Τώρα σε ό,τι με αφορά έχουμε πολλά πράγματα να επιλύσουμε. Πρέπει να ενεργήσουμε από κοινού. Χαίρομαι που άκουσα κυρία ρόζα πως θα γίνει μια συνεδρίαση με το σύνολο του Σώματος των Επιτρόπων αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Θα πρέπει να μπορέσω να ενημερώσω τους επιτρόπους πέραν των διμερών συναντήσεων που έχω με τους επιτρόπους. Θα πρέπει λοιπόν να συναντήσω το σώμα των επιτρόπων για να τους εξηγήσω τι σημαίνει ε, μια κουλτούρα της υπηρεσίας. Λοιπόν, ξέρετε πολύ καλά ότι και στα άλλα θεσμικά όργανα υπάρχουν κάποιες ε, διαφορές, άλλα τμήματα δέχονται την ιδέα να είναι προορατική ε, απέναντι στον πολίτη και να του παρέχουν κάθε υπηρεσία. Υπάρχουν άλλες ε, διευθύνσεις που είναι κάπως επιφυλακτικές, διστακτικές, διότι δεν ε, κατανόησαν απόλυτα περί τίνος πρόκειται. Αυτό λοιπόν θέλω να κάνω με τη βοήθειά σας και γι' αυτό σας ευχαριστώ για την συνεργασία σας. Κυρία Ντέλτσοβα. Σας ευχαριστώ εκ νέου για τα καλά σας λόγια και για το εκτίμηση που δίνεται στον ρόλο του θεσμού δημοσιολαβητή. Ο δημοσιολαβητής εξαρτάται από το κοινοβούλιο. Λοιπόν, η νομιμότητα λοιπόν της οποίας περιβάλλεται ο διαμεσολαβητής οφείλεται στο κοινοβούλιο ακριβώς. Αυτή λοιπόν η νομιμότητα θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντική και του δίνει το ηθικό ανάστημα για να αντιμετωπίσει και να συνεχίσει το έργο του. Πάνω σε αυτό λοιπόν το ηθικό ανάστημα στηρίζομαι. Είναι αυτό είναι κάτι το οποίο μου το παρέχει η στήριξη του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής σας ιδιαίτερα φυσικά ο μηχανισμός της Ένωσης μπορεί να προσφέρει ένα ανθρώπινο πρόσωπο απέναντι στους πολίτες και ελπίζω ακριβώς αυτό να μπορέσω να συνεχίσω να πράττω με την υποστήριξή σας και την ενθάρρυνση σας. Θα ήθελα να επιμείνω στο ότι μπορέσαμε μειώσουμε τον χρόνο διάρκειας των ερευνών αλλά να αναφέρω πως μετά το 2004 είχαμε μια έκρηξη θα έλεγα μια αύξηση της τάξης του 55% των προσφύγων σε σχέση με το 2003 και μας χρειάστηκαν τρία χρόνια περίπου για να μειώσουμε αυτό το άχθος. Ε, τώρα λοιπόν μέσω της ευελιξίας την οποία αναφέρει η κυρία Ρόζα χρησιμοποιώντας ε, πολλές ευέλικτες διαδικασίες όπως ε, την τηλεφωνική συνδιάλεξη η διαδικασία όπως θέλετε. Μπορέσαμε λοιπόν να περιορίσουμε τον χρόνο ολοκλήρωσης της διαδικασίας σε λιγότερο από ένα χρόνο. Αυτό δείχνει πως ε, εφαρμόζουμε και εμείς ως δημοσιολογητές ε, την ε, κουλτούρα και την νεοτροπία της υπηρεσίας και της παροχής υπηρεσιών. Αυτό που είναι θεμελιώδες λοιπόν είναι να επωφελθούμε δύο πραγμάτων. Πρώτον το ότι υπάρχει ένας χάρτης δεσμευτικός και ως εκ τούτου του άρθρου 41 και η αρχή της χρηστής διαχείρισης είναι ένα θεμελιώδες δικαίωμα μετά από τη θέση της ισχυριστικής της αγώνας και να προσπαθήσουμε να προχωρήσουμε σε ένα πεδίο που είναι ιδιαίτερα δύσκολο στο πλαίσιο του όρου fair που είναι πολύ δύσκολο να ερμηνευτεί στα γαλλικά δεν πρόκειται ακριβώς για δικαιοσύνη ή για ισότητα αλλά κάτι το ανάμεικτο. Λοιπόν, πώς θα υπάρξει χρηστή διαχείριση πέραν ε, των ε, λειτουργιών των δικαστηρίων, διότι η έννοια του fairness ε, της ισότητας και της δικαιοσύνης είναι οι δύο άξονες θέλω να δράσω και σας ευχαριστώ εκ νέου κυρία σας ευχαριστώ πολύ για τα σχόλιά σας. Θα ήθελα να πω ότι εκτιμώ ιδιαίτερα τόσο εσάς όσο και όλους τους βουλευτές οι οποίοι μας υποστηρίζουν. Κατέγραψα, κατέγραψα το ζήτημα των ε, επιστολών ε, έγκαιρης ε, της, επιστολών όχλησης, αλλά όπως ξέρετε δεν είμαι δικηγόρος και δεν θα ήθελα να ανακατευθώ σε χωράφια τα οποία δεν γνωρίζω σε βάθος. Πάντως ε, θα ήθελα να πω ότι φαντάζομαι το εξή. Το, το δικαστήριο και οι ε, συνθήκες αναγνωρίζουν τη διακριτικότητα της ε, Κομισιόν για την αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων και αυτό αναγνωρίζεται σε μια ευρύτερη, με την ευρύτερη έννοια και όπου η άσκηση αυτής της ε, διακριτικής μεταχείρισης θα μπορούσε να οδηγήσει σε κάποιες αυθαιρεσίες. Δηλαδή με λίγα λόγια εγώ δεν θα εμπλακώ σε μια τέτοια υπόθεση κατά πόσον δηλαδή η Κομισιόν θα πρέπει να αποστείλει μια υπόθεση στο δικαστήριο ή αν θα την κλείσει, θα την αρχιοθετήσει ή όχι. Εγώ θα παρέμβω στην περίπτωση όπου η Κομισιόν δεν ενεργεί και δεν αποφασίζει. Και έτσι και με αυτόν τον τρόπο τη διακριτική της ευχαίρεια. Ε, σε αυτό ε, συνέβη στο παρελθόν σε αρκετές περιπτώσεις ε, και τελικά αποφάσισε και το φυσικά το τι πώς θα αποφασίσει αυτό ναι εμπίπτει στο πλαίσιο της διακριτικής της και ήθελα να πω ότι θα επανέλθω στο ζήτημα που θέσατε για το ζήτημα των επιστολών όχλησης αλλά θα επανέλθω όταν θα γνωρίζω κάπως περισσότερα περί αυτού. Ευχαριστώ κύριε Κάσμαν για τις παρατηρήσεις σας. Θα ήθελα να προτείνω ότι το θέμα το, του, του ε, της αμαρτίας είναι και ζήτημα κοσμικό. Να, να πω πως ως άθεος ε, αυτό δεν ε, μου δίνει ιδιαίτερη δεν μου δίνει ιδιαίτερη παρηγοριά. Τώρα, σχετικά με το ερώτημά σας κύριε Κάσμαν, να σας πω για μια ακόμα φορά ότι αναπόφευκτα, δεδομένου του μεγέθους των θεσμικών οργάνων, πολλές ε, ε, προσφυγές που γίνονται για την μη παροχή εγγράφων ε, προέρχονται από την, μάλλον ότι στην Κομισιόν. 56-60% είναι οι περισσότερες προσφύγες και επειδή ε, τα δύο τρίτα των ε, δημοσίων υπαλλήλων ε, στα θεσμικό οργάνων εργάζονται στην Κομισιόν, άρα τα περισσότερες προσφυγές και παράπονα προέρχονται από την σχέση του κοινού με την Κομισιόν. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχει ότι την ευθύνη τη φέρνει η Κομισιόν, απλά έχει πιο, πολλού έχει πιο πολλούς υπαλλήλους, πιο πολλά έγγραφα κλπ. Γι' αυτό και το 56 με 60% προέρχονται από, το, από την Κομισιόν, από την ΕΠΣΟ γύρω στο 10%, το Συμβούλιο 2%. Αυτά είναι χοντρικά τα ποσοστά σχετικά με την πρόσβαση στα έγγραφα. Ε, συνεργάζομαι πολύ, μάλλον συνεργάζεται πολύ η Κομισιόν ε, μαζί μου και όπως και τα περισσότερα θεσμικά όργανα δείχνουν κάποιες ε, εσωτερικές διαφωνίες. Δεν είναι ενιαία σώματα. Ως εκ τούτου υπάρχουν ε, κάποιοι θύλακες που είναι υπέρ της συνεργασίας ε, με τον ε, διαμεσολαβητή και επιτρέπουν την πρόσβαση, αλλά υπάρχουν και άλλα, άλλοι θύλακες οι οποίοι είναι λιγότερο δεκτικοί σε κάτι τέτοιο. Και με τον κύριο Ρομέρο προσπαθήσαμε να βελτιώσουμε την κατάσταση. Και ο Ρομπέρο έλαβε καθήκοντα πέρυσι. Όπως σας είπα, σε μερικές φορές υπάρχουν επιφυλάξεις, τη σταγμή και σε άλλες, άλλες φορές υπάρχει άρνηση. Τώρα με το Κοινοβούλιο η συνεργασία μας είναι πολύ καλή σε ό,τι φορά την πρόσβαση στα έγγραφα ε, πέρυσι μπόρεσα να επιλύσω κάποιες ε, τέτοιες υποθέσεις ε, και δεν θα ήθελα να αναφέρω εδώ στην Επιτροπή σας ότι υπήρξαν στιγμές στο παρελθόν ειδικά σε ό,τι αφορά τα οικονομικά των βουλευτών που οδήγησαν σε τριβές της ε, Επιτροπής με τον διαμεσολαβητή. Αυτό έχει να συμβεί μερικά χρόνια τώρα και όπως είπα κύριε Τάσμαν, όσο ε, έχει το καθεστώς του διαμεσολαβητή και της συνθήκης, ο διαμεσολαβητής ε, μπορεί να ασκεί τα καθήκοντά του και απέναντι στο Κοινοβούλιο και πραγματικά το καταστατικό μου αλλά και ε, συνθήκες που είναι τη δυνατότητα να ασκήσω το, το, τα καθήκοντά μου σύμφωνα με τον νόμο και ελπίζω αυτό να μην αλλάξει και αυτό προς όφελος της διαφάνειας αλλά και των ιστορικών διαδικασιών του Κοινοβουλίου. Τώρα για το Συμβούλιο, σας πω έχουμε τα λιγότερες προσφυγές σε ό,τι φορά την πρόσβαση στα έγγραφα. Η αναθεώρηση του καταστατικού πέρυσι προέβλεψε μια ενίσχυση της έννοιας ε, των ε, απορρίτων και εμπιστευτικών εγγράφων. Ε, αυτά, αυτά τα έγγραφα αφορούν ιδιαίτερα στο Συμβούλιο, αλλά έχουμε τη δυνατότητα τώρα να έχουμε πρόσβαση στα χαμηλότερο χαρακτηρισμό, αν θέλετε, στα restricted, και είμαι γνώμων στην Σουηδική Προεδρία που μου διευκόλυνε την πρόσβαση στα έγγραφα αυτά τα restricted και μέχρι σήμερα μπορέσαμε να βρούμε ε, τρόπο για να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση αυτή των ε, διαβασισμένων εγγράφων. Κυρία Μπαζέσκου, ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Πολύ χαίρομαι για τα καλά λόγια για τον διαμεσολαβητή, όπως και για τις επικρίσεις που μας βοηθούν να κάνουμε καλύτερα τη δουλειά. Για το ECI, με την άδειά σας θα μιλήσω για το ECI σε συνδυασμό με τις παρατηρήσεις του κυρίου Χέφνερ για να δώσω μια ενιαία απάντηση αν μου επιτρέπετε γιατί έχουν τεθεί πολλές ερωτήσεις και πρέπει να ε, ομαδοποιήσω και λίγο. Η κυρία Σντανόγκα, εδώ δύο απαντήσεις οφείλω. Αντιλαμβάνεστε ότι εξορισμό ορισμού διαμεσολαβητής δεν εξουσιοδοτείται να ασχοληθεί με νέα νομοθεσία. Αυτό είναι το δικό σας κατεξοχήν κοινοβουλευτικό έργο. Εγώ θα πρέπει να παρεμβαίνω αφού εγκρίνετε εσείς την νομοθεσία που θα τίθεται σε εφαρμογή και θα κρίνουμε πια την εφαρμογή του, πόσο καλή ή κακή είναι. Αυτό που κάνω εγώ είναι να παρακολουθώ εκ του σύνεγγης και ε, βλέπω τις προσπάθειες, νομοθετικές προσπάθειες σε σχέση με την καλή διαχείριση, τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών. Αυτό είναι το έργο του διαμεσολαβητή και λόγω της εξαιρετικής ε, σχέσης με την Επιτροπή σας ενημερώνω το Κοινοβούλιο μέσα από την Επιτροπή Αναφορών ή Πολιτικών Ελευθεριών ή Συνταγματικών Υποθέσεων και κοινοποιώ τις απόψεις μου εσείς ε, κυρίαρχα θα αποφασίσετε τι θα κάνετε και όταν εγκρίνετε τον νόμο θα δω πώς μπορώ εγώ να κινηθώ σε επίπεδο εφαρμογής του. Τώρα, για το συγκεκριμένο σας ερώτημα, σε ό,τι αφορά την ενδεχόμενη δημιουργία διοικητικού δικαίου, αυτό προβλέπεται στο άρθρο 298 της συνθήκης. Και η θέση μου είναι ότι και οι προκάτοχοί μου και εγώ προσπαθήσαμε να το προωθήσουμε αυτό και διαπιστώσαμε ότι τα θεσμικά όργανα ακόμα δεν είναι απόλυτα έτοιμα να κινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση. Έθεσα το θέμα στην κυρία Βάλστρομ όταν ήταν αντιπρόεδρος της Επιτροπής και εκείνη επίσης ήθελε πολύ να δοθεί συνέχεια στο θέμα. Όμως ε, φάνηκε ότι σε τελευταία ανάλυση η θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ότι εμείς προβλέπουμε την δυνατότητα να συμβεί κάτι τέτοιο στο μέλλον, όμως ακόμη δεν έχουμε φτάσει στο σημείο αυτό. Προφανώς ε, πρόκειται για έναν ακόμη τομέα όπου θα πρέπει ε, να υπάρξει ε, νομοθετική πρωτοβουλία. Τώρα, να προσθέσω κάτι που ίσως είναι πιο αμφιλεγόμενο, αλλά απευθύνομαι σε μια επιτροπή που είναι πολύ κοντά στο διαμεσολαβητή. Η δημιουργία ενιαίου δικαίου θα επέφερε πολλά ωφέλη στους πολίτες, διότι θα υπήρχε μια σειρά κανόνων ε, για να χρησιμοποιούν. Κατόπιν τούτου, ο ιδιαίτερος ρόλος του διαμεσολαβητή είναι να μπορεί να εργάζεται αυτό που θα έλεγα πέραν του νόμου, όχι εκτός νόμου, αλλά πέραν του νόμου. συνήθως τους διασκεδάζω τους ε, νομικούς συνομιλητές μου όταν τους λέω ότι υπάρχει ε, ζωή πέραν των νομικών χωρίς να θέλω να πω ότι ε, είναι πέραν του νόμου. Υπάρχει όμως μία διαφορά μεταξύ της νομιμότητας που οριοθετεί το ελάχιστο απαιτούμενο από τον νόμο και η καλή διαχείριση που θα πρέπει να πάει πέραν του νόμου και οι απαιτήσει μιας δημόσιας διοίκησης ε, που λέει ότι δεν, δεν, δεν μπορεί να περιορίζεται στο ότι δεν έχει παραβιαστεί ο νόμος. Η μη παραβίαση από τη μία και το όριο δηλαδή της καλής διακυβέρνησης είναι το πεδίο που κινείται ο διαμεσολαβητής διότι πολλές φορές ε, νομικά μπορεί να περιορίζεται η διακριτική ευχέρεια του διαμεσολαβητή που κινείται ακριβώς αυτό το όριο μεταξύ νόμου και καλής διακυβέρνησης. Όμως είμαι πεπισμένος ότι ο διαμεσολαβητής πάντα θα μπορεί να δρά πέρα, πέραν των στενών ορίων της νομιμότητας για την καλή διαχείριση και την βοήθεια και υποστήριξη των πολιτών. Από αυτή την έννοια, αν υπάρχει νόμος, ε, που θα προάγει την καλή διακυβέρνηση. Αυτό είναι υπέρ και του διαμεσολαβητή και των πολιτών, αλλά σε τελευταία ανάλυση οι νομοθέτες, η νομοθετική αρχή εσείς θα αποφασίσετε. Τώρα, να απαντήσω και στον ε, κυρία Μπαζέσκου και τον κύριο Χέφνερ. Καταρχήν κύριε Χέφνερ, Είμαι στη, απόλυτα στη διάθεσή σας και ευχαριστώ για την προσφορά συνεργασίας. Πάντοτε άμεσα και με ευχαρίστηση απαντώ σε προσκλήσεις ε, του Κοινοβουλίου και των Επιτροπών του ε, και των πολιτών για συνεργασία προς το συμφέρον των πολιτών. Σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στα έγγραφα, με χαρά θα βοηθήσω την Συνταγματική Επιτροπή για να γίνει κάτι περισσότερο. Ως Έλλην να σας συγχαρώ και για την ε, άψογη αυτή ε, τελική σας παρέμβαση. Ναι, ήταν η κυρία Καγιατεμέκη. Αλλά μπορώ να έρθω στην Επιτροπή ε, Ευχαριστώ, αν με καλέσετε, όπως έκανα και στο παρελθόν, για να συζητήσουμε. Τώρα, για την ε, Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών, εγώ έχω παρουσιάσει και έχω εκθέσει τις απόψεις μου από αυτού πολλές φορές και κοινοποίησα ε, το θέμα αυτό της δημόσιας ακρόασης, ε, τη διαβούλευσης ε, που πρόθεσε και η Κομισιόν. Είναι ένα καλό εργαλείο που πρέπει να παρακολουθείτε προσεκτικά για να αποφεύγονται πιθανές απογοητεύσεις των πολιτών. Εγώ πιστεύω και νομίζω ότι και πολλοί άλλοι το πιστεύουν αυτό ότι ένα εκατομμύριο υπογραφές ε, στο διαδίκτυο, στην εποχή του διαδικτύου δεν είναι μεγάλο εμπόδιο Ιδιαίτερα οι καλά οργανωμένοι φορείς που έχουν υποδομή εύκολα συγκεντρώνουν ένα εκατομμύριο υπογραφές. Άρα λοιπόν είναι ακόμα πιο σημαντικό να διασφαλίζουν τα θεσμικά όργανα ότι η πρωτοβουλία των Ευρωπαίων πολιτών θα ε, πραγματοποιείται πολύ προσεκτικά ευθύς εξ αρχής. Και αυτό σημαίνει, και το λέω σε μια κοινοβουλευτική επιτροπή, ότι η πρωτοβουλία των πολιτών θα συντονίζεται πολύ από την Κομισιόν, αλλά δεν θα είναι ένας μηχανισμός μόνο προς όφελος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα είναι μηχανισμός που θα επιτρέπει και στο Κοινοβούλιο να παρεμβαίνει με τρόπο ουσιαστικό διασφαλίζοντας ότι οι διατάξεις της συνθήκης της Λισαβόνας που προβλέπουν ε, καλύτερο διάλογο, περισσότερες επαφές μεταξύ αυτού του Κοινοβουλίου και των Εθνικών Κοινοβουλίων και συμμετοχή και διάλογο σε τελευταία ανάλυση με τους πολίτες διασφαλίζονται από αυτό το φορέα επίσης και η πολίτες είναι οι διπλά ωφελούμενοι αποδέκτες αυτών των πρωτοβουλειών. Έχοντας αυτά κατά νουν, υπέβαλα τη σχετική πρόταση και ευχαρίστως να σας την στείλω αν δεν την έχετε. Η πρόταση προβλέπει καταμερισμό εργασίας μεταξύ Κοινοβουλίου και Διαμεσολαβητή για την διασφάλιση της διαδικαστικής ε, ακαιρεότητας του ACI, Θα μπορεί δηλαδή σε νομικά θέματα να αποφαίνεται ο διαμεσολαβητής για τις διαδικασίες. Το παραδεκτό, την καταχώρηση, γιατί σίγουρα θα υπάρχουν προσφυγές προς τον διαμεσολαβητή, όπως έρχονται και στην Επιτροπή Αναφορών, για τα διαδικαστικά. Οπότε ο διαμεσολαβητής θα αποφαίνεται επί των νομικών διαδικαστικών θεμάτων, αλλά εγώ είπα ότι θα πρέπει και το Κοινοβούλιο να εξετάζει τα, την ουσία, την πολιτική ουσία που αναφέρεται στο περιεχόμενο αυτών των πρωτοβουλειών, ώστε να μην υπάρξει περίπτωση κάποια στιγμή μετά τη συλλογή, συγκέντρωση ενός εκατομμυρίου υπογραφών να πει Κομισιόν απαράδεκτο και οι πολίτες να νιώθουν απογοήτευση ε, αν όχι και ότι εξαπατήθηκαν. Η πρόταση προβλέπει συγκεκριμένο ρόλο για το Κοινοβούλιο λοιπόν στον τομέα της ε, επανεξέτασης ε, της ουσίας των πρωτοβουλειών και του περιεχομένου τους, ώστε να μπορέσει η Κομισιόν να ασκήσει την εντολή της στα πλαίσια του κανονισμού προς όφελος όλων των πολιτών. Και είμαι στη διάθεσή σας βεβαίως ε, να έρθω στην Επιτροπή σας ή σε οποιαδήποτε άλλη κοινοβουλευτική επιτροπή για να παρουσιάσω τις απόψεις μου, όποτε το θελήσετε. Ελπίζω να απάντησα στην ερώτησή σας. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Δία Μεσολαβητά Διαμαντούρο. Πολλή δουλειά έχει γίνει, αλλά μην ε, αρκεστείτε σε αυτά, να είστε απαιτητικός, διότι έχετε πολλά ακόμα να κάνετε. Θα σας δώσω το λόγο αμέσως για την ε, παρουσίαση της ειδικής έκθεσης ε, και θα δώσω και το λόγο στην κυρία Παλιαδέλη, που είναι η συγκητριά μας. Ζητώ να μην μακρυγορίζετε, διότι έχουμε και άλλα δύο θέματα να ολοκληρώσουμε πριν από τις 12.30. Ευχαριστώ. Θα είμαι πιο σύντομος παρουσιάζοντας αυτήν την ε, ειδική έκθεση διότι εξ ορισμού είναι μια έκθεση που δεν είναι τόσο μακροσκελής όσο η έκθεση που αφορά τις δραστηριότητες μια ολόκληρης χρονιάς. Προέδρε, αγαπητά μέλη, με αυτή την ευκαιρία να σα κάνω μια σύντομη εισήγηση όσον αφορά αυτή την ε, πάγια συμφωνία μα. Ότι δηλαδή θα έρχομαι εδώ οποτεδήποτε έχουμε κάποια έκθεση την οποία πρέπει να βάλουμε στο Κοινοβούλιο. Και θα έρχομαι στην Επιτροπή. Και ε, αυτή, ε, αυτό είναι το, τελευταίο καταφύγιο, το, το, το, το, έσχατο όπλο που έχει διαθέσει ο Μεσολαβητή. Όπω σα είπα, δεν έχω τη δύναμη να λαμβάνω νομικά δεσμευτικέ αποφάσει. Όμω αυτό το οποίο μπορώ να κάνω είναι να προβάλλω επιχειρήματα για να στηρίζομαι στην κοινή γνώμη. Και είναι τελικά πάρα πολύ λίγε οι ειδικέ εκθέσει που έχει υποβάλει ο Μισολευτή στο Κοινοβούλιο, ε, δηλαδή 17 τον αριθμό σε 14,5 χρόνια. Αυτό καταδεικνύει το πόσο υπάρχει προσέγγιση συνεργασίας στις περισσότερες περιπτώσεις μεταξύ των θεσμικών οργάνων. Και βέβαια το ιστορικό πλαίσιο, το background είναι το ότι μπορούμε Ακριβώ να υποβάλλουμε μια τέτοια δική έκθεση, ιδίως όταν έχουμε με ένα σχέδιο σύστασης. Το, το, το, το ότι γνωρίζουμε το μπορεί να υπάρξει τέτοια δική έκθεση, αυτό βοηθάει όσον αφορά την συνεργασία των θεσμικών οργάνων, γιατί οι ειδικέ εκθέσει δεν θα πρέπει να είναι κάτι στο οποίο προσφέρουν πάρα πολύ συχνά, όμω θα πρέπει να γίνεται και κάποια σημαντικά ζητήματα, ώστε να μπορέσουμε να πείσουμε ε, τα θεσμικά όργανα για τις θέσεις μας. Και ως όργανο πολιτικό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι κυρίαρχο όσον αφορά αυτές τις ειδικέ εκθέσεις. Όσον αφορά δε τη διαδικασία αλλά και την ουσία της ε, προσέγγισης αλλά και της ενέργειας που αναλαμβάνονται. Παρ' όλα αυτά, ε, ελπίζω ότι όταν έχετε η ώρα της ειδική έκθεσης το Κοινοβούλιο θα πρέπει πάντοτε να, να λαμβάνει υπόψη ότι ε, είναι πάρα πολύ θεμελιώδης δικαίωμα ενός πολίτη η υποβολή των αναφορών. Ε, είναι κάτι το οποίο κατοχυρώνεται με αυτόν τον χάρτη των ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έχει νομική ισχύ δυνάμει συνθήκη τη Λισαβόνα. Και για του λόγου που σα εξήγησα, οι ειδικέ εκθέσει αλλά και η ανταπόκριση του Κοινοβουλίου θεωρούνται ο ακρογωνίο λήθο και θεμέλιο του έργου του διαμεσολαβητή. Τώρα, όσον αφορά την ειδική έκθεση που υπέβαλε στο Κοινοβούλιο στις 24 Δευτέρου είναι στο και αφορούσε την ε, έρευνά μου ε, ε στην υπόθεση 676 του 2008. Διότι δεν συνεργάστηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά την ε, διεκπαιρέωση αυτή τη υπόθεση. Οπότε είχα αυτή την ειδική έκθεση για να μπορέσει να με βοηθήσει το Κοινοβούλιο στο μέλλον και έτσι η Κομισιόν να τηρεί την υποχρέωση συνεργασίας. Το ιστορικό πλαίσιο έχει ότι τον Μάρτιο του 2007 μια μη κυβερνητική οργάνωση η οποία ενεργούσε ε, για θέματα περιβάλλοντος ζήτησε προσβασιμότητα ε, σε κάποια έγγραφα δυνάμει του οργανισμού 1049 του 2001 και ε, αφορούσε τον, τον έλεγχο εκ μέρους της Κομισιόν των εκπομπών διοξείδου του άνθρακος επί των αυτοκινητοβιομηχανιών και τελικά 15 από τις 18 επιστολές που είχε αναποσταλεί στον τότε αρμόδιο Κίντερ Φερχόγεν ε, αυτά κοινοποιήθηκαν. Όμως είχαμε τρεις επιστολές της Πόρσε και θεωρήθηκε ότι είναι διαφορετημένες αυτές οι επιστολές και ότι πρόκειται να παραβλαβούν τα εμπορικά συμφέροντα της ε, της εταιρείας. Ε, οπότε στράφει αυτή η οργάνωση στον διαμεσολαβητή και το 2008 ε, προσφύγαμε και καταφύγαμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταλήξαμε ε, να ολοκληρώσουμε τη δικασία στις 27 Δεκάτου 2008 και καταλήξαμε στο ότι είχε αρνηθεί προσβασιμότητα εκ μέρου τη Κομισιόν και κάναμε ένα σχέδιο σύσταση προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θα πρέπει να δώσει πρόσβαση σε αυτές τις επιστολές ε, εν όλο ή εν μέρη. του άρθρου 6, συγγνώμη, το άρθρο 3 παράγραφος 6 σε σχέση με τον κανονισμό λειτουργίας που έγινε το Κοινοβούλιο και τότε έστειλε μια επιστολή λεπτομερή Ευρωπαϊκή Επιτροπή 31 πρώτου του 2009. Ε, δεν απάντησε στην υποστολή μου αυτήν η Κομισιόν και ζητήθηκε παράταση προθεσμίας στις 30 ε, Ιανουαρίου μετά ζητήθηκε αυτό και τέλος Φεβρουαρίου και στις 26 ε, Μαρτίου και άλλη παράταση και ζήτησαν και άλλη παράταση στις 29 Τετάρτου του 2009. Επίσης ζητήσανε για άλλη παράταση στις 29 Πέμπτου του 2009 και ακόμα μια φορά στις 26 Έκτου του 2009. δινόταν κάθε φορά η προθεσμία και τελικά απίφθηνα του 2009 μια επιστολή και έλεγα ότι θα πρέπει να μου πούνε ακριβώς γιατί η σύνταξη μιας ε, σύστασης παίρνει τόσο πολύ χρόνο και γιατί ζητήθηκαν έξι παρατάσεις μιας ήδη άνετης προθεσμίας. Αμέσως απήντησε η Κομισιόν στην επιστολή μου στις 17 Εβδόμου και είπε ότι δεν είναι η θέση να δώσει μια αιτιολογημένη απάντηση ε, διότι ακόμα βρίσκεται σε διαβουλεύσεις με την Πόρσε. Στις 30 Σεπτεμβρίου 2009, 10 μήνες μετά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μου είπε ότι αποφάσισε να επιτρέψει την πρόσβαση σε αυτές τις επιστολές εν μέρη. Και ε, αποφάσισαν να, να, το πούνε αυτό και στην Πόρσε στις 27 του 2009 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξήγησε ότι η απόφαση για ενημέρωση της Κομισιόν πάει για να μεταφραστεί στα γερμανικά και αρχάς Νοεμβρίου πρόκειται να πάει στην εταιρεία. Σε 9-10 έστειλα και άλλη μια επιστολή και ζήτησα ένα αντίγραφο αυτή τη ειδοποίηση προ την Πόρσε, ούτω ώστε να με ενημερώσουν για το τι γίνεται όσον αφορά την πρόσβαση αυτή τη επιστολή. Στι 4 2009 οι Κομισιόν μα ενημέρωσαν τηλεφωνικά ότι άμεσα θα μας διαβάσουν, θα διαβάσουν συγγνώμη, την επιστολή στην Πόρσε και, και, την, ε, και το αντίγραφο. Στις 20 Φεβρουαρίου 2010 ακόμα δεν είχα λάβει τίποτα. Ούτε αντίγραφο τη ειδοποίηση, ούτε ενημέρωση για το τι έγινε με την πρόσβαση στα έγγραφα. Μόλι ε, εγκαταστάθηκε ανέβη καθήκοντα νέα επιτροπή, τότε η Κομισιόν όντω επέτρεψε την προσβασιμότητα στα έγγραφα. Αυτό όμω έγινε με καθυστέρηση 15 μηνών μετά το σχέδιο της σύστασης και όχι ε, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας ε, που λέει ότι πρέπει να γίνει σε τρει μήνες και σύμφωνα με το άρθρο 200 της συνθήκης. Οπότε, εγώ απίθανα επιστολή και είπα γιατί δεν το έκαναν αυτό όποτε έπρεπε και Είχε εξηγήσει η Κομισιόν που τρέχονταν σε επαφή μαζί μα ότι δεν μπόρεσε να συμμορφωθεί με αυτή την προθεσμία των τριών μηνών γιατί συνεχιζόντουσαν οι συνεννοήσει με την Πόρση όσον αφορά ε, την ε, αποκάλυψη, την, την, την προσβασιμότητα σε αυτέ τι ε, επιστολέ. Και σαν επιχειρήματα προέταξε η Κομισιόν ότι πρώτα-πρώτα σε αυτέ τι διαπραγματεύσει με την Πόρση θα υπήρχε κάποιο ε, θετικό αποτέλεσμα όσον αφορά την προσβασιμότητα σε επιστολές και ότι θα έπρεπε να μπορέσει να έχει υπόψη αρκετό χρόνο, ούτως ώστε να μπορεί να προσφύγει κατά της Κομισιόν, κατά της απόφασης ε, αποκάλυψης των επιστολών. Όσον αφορά το πρώτο επιχείρημα. Έχουμε τώρα το 4 παράγωγος 4 του κανονισμού 1049 και προβλέπει ότι θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ορίσει για κάθε ε, τρίτο μία προθεσμία όσον αφορά την, ε, την, την την απάντηση για κάποιο έγγραφο. Ε, θα πρέπει επομένω να τηρεί αυτό το οποίο θεσπίζει η Διεπιτροπή. Σε αυτό το δεύτερο ε, επιχείρημα, έχουμε να πούμε ότι το να επιτραπεί στην ε, Πόρσε να ασκήσει τα νόμια δικαιώματά τη δεν δικαιολογεί αυτή την μεγάλη καθυστέρηση. Άρα δεν χρειαζόταν 15 μήνες για να φτάσει στην κοινοποίηση αυτή, στην ενημέρωση αυτή. Επίση υπάρχει αρχή τη ειλικρινού συνεργασία που είναι κατοχυρώνεται στην ομολογία, αλλά αυτό προβλέπει τώρα το 4 3 τη Συνήθεια Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με το οποίο τα θεσμικά όργανα υποχρεούνται να συνεργάζονται καλόπιστα με το ένα με το άλλο. Και σας παραπέμπω και στο άρθρο 13 παράγραφος 2 της νέας συνθήκης. Επομένως, καταλήγω στο ότι με αυτή τη καθυστέρηση των 15 μηνών όσον αφορά το σχέδιο σύσταση και διότι τελικά δεν ενημερώθηκε η Πόρσε σε σχέση με το άνοιγμα των επιστολών παραβιάστηκε εκ μέρους της Επιτροπής η υποχρέωσή της να συνεργάζεται ειλικρινά και καλόπιστα. Κατά αυτή την έρευνα θεώρησε ότι υπάρχουν φαινόμενα εδώ κακοδιοίκησης και είχε κάθε φορά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την ευκαιρία να επανορθώσει. Και αυτόν τον τρόπο υπονομεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την εμπιστοσύνη των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά και τη δυνατότητας του Διαμεσολαβητή να εποπτεύει το θεσμικά όργανα και τη την Επιτροπή. Και επίσης αυτό αντιβαίνει στην αρχή του κράτους δικαίου. Το ίδιο αφορά και σε αυτές όλες τις ε, παρατάσεις. Τώρα μιλάμε για καθυστέρηση ενό έτου αντί για του τρει μήνε που προβλέπει το Κοινοβούλιο σαν προθεσμία. Και άρα θα πρέπει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να λάβει υπόψη αυτή την ειδική έκθεση και θα πρέπει το Κοινοβούλιο να ζητήσει από την Κομισιόν πρώτα-πρώτα να αναγνωρίσει ότι αυτή η υπερβολική καθυστέρηση στο να ανταποκριθεί στα αιτήματα του διαμεσολαβητή αποτελεί παραβίαση του, της υποχρέωσης ε, ειλικρινούς συνεργασίας όπως προβλέπει η συνθήκη και δεύτερον να ζητηθεί, να δεσμευθεί προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Κομισιόν ότι θα τηρεί τις υποχρεώσεις της στο μέλλον. Euh, Ευχαριστώ. Οι πολίτες μας θα πρέπει πάντα να έχουν εμπιστοσύνη στα όργανα μας. Να δώσω το λόγο στην κυρία Παλιαδέλη που είναι η συγκητρία εισηγήτρια, υπήρξα εισηγήτρια με απόλυτα... Ε, ε, ήταν εξαιρετική τιμή ότι ήμουν εισηγήτρια για την εισήγηση για, την πενταετία του κυρίου Διαμαντούρη στην προηγούμενη θητεία του. Απλώς έχω κάνει μια ερώτηση που αφορά στο ίδιο θέμα, <laughs> την οποία θα την απευθύνω στη συνέχεια. Επομένω, γράψτε με στον κατάλογο των ομιλητών σα παρακαλω Θέλω να κάνω μια ερώτηση στον ε, κύριο Διαμαντούρο και μια ερώτηση στην Επιτροπή. Η ερώτηση στον κύριο Διαμαντούρο είναι αν έλαβε στη συνέχεια ε, τα, τις επιστολές προς την Πόρσε ε, που τόσο καιρό προσπαθούσε να λάβει και μία ερώτηση προς την Επιτροπή η οποία σε ερώτηση δική μου γραπτή και του κυρίου Αρσένη από κοινού, μία ερώτηση ε, του κ. Αρσένη και δική μου, με αφορμή αυτή την καθυστέρηση, την υπόθεση με την Πόρσε, η Επιτροπή μόλις πρόσφατα μου απάντησε με αυτόν εδώ τον απαράδεκτο τρόπο, λέγοντας ότι μας παραπέμπει στην απάντηση σε μια προγενέστερη ερώτηση που είχε κάνει ένας άλλος ε, συνάδελφος, ένα άλλο μέλος του Ευρωπαϊκού ε, Κοινοβουλίου. Η ερώτηση αυτή, την οποία έψαξα να βρω, του συναδέλφου κάνει διαφορετικά ερωτήματα ε, και δεν απαντάει εν τέλει στα δικά μου ερωτήματα, του κύριου Αρσένη και τα δικά μου. Θεωρώ ότι αυτή η διατύπωση από τον κύριο Μπαρόσο, η, η, απάντηση λέει, απάντηση του κυρίου Μπαρόσο εξ ονόματος της Επιτροπής 28 Τετάρτου 2010, λέει ως εξής. Η Επιτροπή παραπέμπει τα αξιότιμα μέλη, εννοεί τον κύριο Αρσένη και εμένα, στην απάντησή της στη γραπτή ερώτηση τάδε του κυρίου Μποργκέτσιο. Πρώτον, η απάντηση δεν ισχύει και για τη δική μου ερώτηση και του κυρίου Αρσένη. Και δεύτερον, ομολογώ ότι δεν έχω υποστεί ποτέ μεγαλύτερη ταπείνωση αποδεχόμενη αυτήν εδώ την έκφραση ως απάντηση του, της Επιτροπής απέναντι σε ένα μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Περιμένω λοιπόν απάντηση και για αυτό το πράγμα. Ευχαριστώ πολύ. Je vais donner la parole à Madame Auken. Så tror jeg, jeg vil tale dansk. For at... Θα μιλήσω την μητρική μου γλώσσα, την δανική. για να διατηρήσω και τους ε, διερμηνείς εφόρμα να μην ξεχνούν την ε, δανεική γλώσσα. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να πω πως ευχαριστώ εκ βάθους καρδίας ε, τον εισηγητή για την ειδική αυτή έκθεσή του που έχει ιδιαίτερη σημασία. Σπανίζει να παρατηρούμε τέτοια φαινόμενα απέναντι όχι μόνο στους ε, πολίτες αλλά και απέναντι στον ε, διαμεσολαβητή αλλά και όλων ημών εξάλλου. Η όλη διαδικασία ήταν ε, πολύ ενδιαφέρουσα, υποδειγματική θα έλεγα και έχω μια ερώτηση να θέσω. Γιατί η σύμβαση όρους δεν αναφέρεται στην περίπτωση αυτή γιατί η Κομισιόν κατά την άποψή μου θέλησε να υποστηρίξει ένα, μια μεγάλη βιομηχανία κατά των πολιτών και κατά του περιβάλλοντος. Θα έπρεπε λοιπόν εδώ να υπάρχουν επιβαρυντικά στοιχεία. Αυτό λοιπόν πιστεύω ότι μας αφορά όλους διότι είμαστε όλοι υποχρεωμένοι να τηρούμε την σύμβαση Άρους. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι θα έπρεπε να αναφέρεται στα κείμενα και να πω επίσης στην κυρία Παλιαδέλη πως αυτό που είπες προλίγου θα πρέπει να συμπεριληφθεί διότι είναι απαράδεκτο να λαμβάνονται τέτοιου είδους απαντήσεις. Πρώτα απ' όλα δεν απάντησαν άμεσα, είχαν όλο τον χρόνο στη διάθεσή τους προκειμένου να το σκεφτούν το ζήτημα. Άρα η Κομισιόν Ε, στην περίπτωση αυτή δεν ε, είναι η μοναδική που, ε, που κατηγορείται εδώ. Εμεί θα πρέπει να αντιδράσουμε, διότι είναι πραγματικά υποδειγματικό αυτό το οποίο συνέβη. Θα ήθελα να ευχαριστώ τη συνάδελφο για τα όσα είπε, αλλά και αυτά που είπε ο Δημοσιολογητή. Να δώσω το λόγο στον κύριο Εθνάρχο και να ζητήσω να είστε ε, Μετά δεν έχουμε χρόνο να μιλήσει κάποιος άλλος. Ζήτησα το λόγο γιατί έχει γερμανικό υπόβαθρο η περίπτωση αυτή και θα μιλήσω και γερμανικά γι' αυτό. Δύο ερωτήσεις. Πρώτον, μιλήσατε ξεκάθαρα για την ε, υπονόμευση της εμπιστοσύνης. Πώς μπορεί αυτή να επανικοδομηθεί ή για να το πω αλλιώ, αν ένα πολίτη που ως επιτοπλίστων δεν διαθέτει μηχανισμό από πίσω του, είναι μόνος του. Αν χάσει α πούμε, μια προθεσμία θα το πληρώσει ακριβά. Και ε, δεν θα συνεπικουρηθεί από τον νόμο γιατί έχασε την προθεσμία. Ε, εδώ πολλές φορές δεν έχουν τηρηθεί προθεσμίες. Με απασχολεί λοιπόν το ερώτημα πώς θα ξανακερδίσουμε την εμπιστοσύνη ε, του πολίτη, ότι δηλαδή τον παίρνουν στα σοβαρά. Αυτό είναι το ένα που με απασχολεί. Και το άλλο, αν δούμε τα θέματα και πέρα από τα νομικά, όλοι ξέρουμε ότι η Πόρσε, γιατί τότε το θέμα ήταν ο περιορισμός των εκπομπών αυτοκινήτων και η Πόρσε στην Ευρώπη είναι ο κατασκευαστής με τα, τις υψηλότερες εκπομπές. Το έτος που έγινε η ανταλλαγή επιστολών, η Πόρσε ταυτόχρονα ήταν και από τους πιο επιτυχημένους και πιο κερδοφόρους κατασκευαστές. Οπότε μπορεί κανείς να φανταστεί ότι η Πόρσε δεν ενδιαφερόταν και πάρα πολύ για τις ρυθμίσεις που συζητούνταν. Ταυτόχρονα, ο Επίτροπος Βιομηχανίας προέρχεται από τη χώρα που έχει την έδρα της η Πόρσε και υπήρξε μια ανταλλαγή επιστολών και κατάλαβα ότι αυτό ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Αν κατάλαβα καλά, η Κομισιόν δημοσίευσε ε, το το κομμάτι όπου είχε αλληλογραφία ο Επίτροπος Βιομηχανίας με κατασκευαστές Γάλλους ή Ισπανούς, αλλά η αλληλογραφία με τον κατασκευαστή με τις υψηλότερες ε, εκπομπές που είναι από τη χώρα του Επιτρόπου ε, και αυτό δεν αναφέρθηκε. Άρα λοιπόν δεν πρόκειται μόνο για κακοδιοίκηση, για κάποια παράληψη. Δημιουργείται δηλαδή στους πολίτες ή η εντύπωση ότι δεν αντιμετωπίζονται όλοι επίσης όρισε. Και ίσως και το εθνικό υπόβαθρο και ε, η προέλευση του Επιτρόπου ε, κατά την άσκηση του αξιώματός του παίζει ενδεχομένως ρόλο. Ευχαριστώ να δώσω λόγο κύριο Διαμαντούρο και να σας ζητήσω να είστε λακωνικός. Ευχαριστώ. Θα απαντήσω στην ερώτηση της κυρίας Παλιαδέλη και θα απαντήσω στην ελληνική. Παλιαδέλη, I obviously have certain limitations, I, gladly accept them. Um, ε, ε, δέχομαι. Ε, ένας άνθρωπος πρέπει να ξέρει τους περιορισμούς και τα όρια του και εγώ τα δέχομαι τα δικά μου. δεν μπορώ προφανώς εγώ να τοποθετηθώ και δεν με ρωτήσατε να τοποθετηθώ στο θέμα το οποίο απευθύνεται απευθείας στην Επιτροπή. εγώ μπορώ να σας απαντήσω ότι τελικά, η, να, το, να το πω ως Η υπόθεση η οποία αφορούσε τις επιστολές είναι διαφορετική από την ειδική έκθεση η οποία εστάλει στο Κοινοβούλιο. Η υπόθεση με τις επιστολές δεν έχει κλείσει. Είναι ακόμα ανοιχτή. Διότι μετά την ανάληψη των καθηκόντων του κυρίου Σεφτσοβίτς, οι επιστολές τελικά εστάλησαν και αυτή τη στιγμή πήρα τις επιστολές οι οποίες έχουν, από έχουν απαλληφθεί ορισμένα ονόματα. Τις έχω στείλει στον, στον καταγγέλλοντα πολίτη, στην οργάνωση η οποία είχε προσφύγει σε μένα, για τα δικά της σχόλια. Προς το παρόν δεν έχω πάρει, είμαστε μέσα στα χρονικά όρια, μέσα στα οποία περιμένω να πάρω τα σχόλια του, ε, του αναφερομένου όταν θα έχω τα σχόλια αυτά θα καταλήξω εάν χρειάζεται περαιτέρω έρευνα ή όχι, προκειμένου να κλείσω την υπόθεση. Άρα προς το παρόν έχω πάρει τα γράμματα, όμως η υπόθεση παραμένει ανοιχτή. Η, προφανώς, επαναλαμβάνω, το, η ειδική έκθεση είναι απόρρια αυτής της υπόθεσης, αλλά είναι, αλλά είναι αναλυτικά διακριτή από την υπόθεση αυτή. Uh, Κυρία Όκεν, πολύ το προσεκτικά το σημείο σε αυτό που είπατε. Θα το δούμε. Θα μπορούσαμε να έχουμε συμπεριλάβει και μία αναφορά στη Σύμβαση Άρχους, που είναι σαφής. Γιατί δεν το κάναμε, να σας πω. Για το μόνο λόγο ότι προσπαθούσα να επικεντρωθώ στο συγκεκριμένο θέμα που θεωρούσα σπάνιο. Σπάνιο σπάνια περίπτωση κακοδιοίκησης. Πρέπει να ενημερώσω το Κοινοβούλιο και απαντώ εδώ και στον κύριο Χέφνερ, πρέπει να πω και το επαναλαμβάνω ότι είναι η πρώτη φορά στα χρονικά, στα 15 χρόνια τουλάχιστον, της εργασ... του, του μου, πρώτη φορά σε 33 περιπτώσεις όπου ένιωσε περιορισμό ο διαμεσολαβητής και έλλειψη συνεργασίας και ανοιχτής, ειλικρινούς συνεργασίας. Πολύ λυπάμαι που έγιναν έτσι αυτά όλα και το λέω και την παρουσία της κυρίας Κωνσταρόζα. Ασύνηθες τελείως, αλλά δεν είναι θεμητό οποιοδήποτε θεσμικό όργανο να ε, καθυστερεί, να αναγνωρίσει τα προβλήματα και να καθυστερεί να απαντήσει ε, σε μια σύσταση ε, η οποία αφορά ε, παραδιάσεις και επί 15 μήνες. Προσπαθώ να κρατήσω σύντομη την έκθεση. Το σημείο όμως αυτό που είπατε για μελλοντική χρήση και αναφορά. Κατόπιν τούτου να απαντήσω και στην ερώτηση του κυρίου Χέφνερ στα σχόλιά του. Κύριε Χέφνερ, ο διαμεσολαβητής πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός στο πώς χειρίζεται τα θέματα, ούτω ώστε να διασφαλίζει την ακαιρεότητα της διαδικασίας. Δεν θα επιτρέψω στον εαυτό μου εικασίες σχετικά με τους λόγους γιατί οι επιστολές αυτές δεν μου εδόθησαν νωρίτερα. Το γεγονός ότι δεν μου εδόθησαν είναι ένα περιστατικό κακοδιοίκησης και αυτό το καταγράφω και το λέω και στο Κοινοβούλιο. Επίσης καταγράφω την εκτίμησή μου για το γεγονός ότι όταν ο νέος επίτροπος, όταν η ε, ε, ε, κυρία Σέκοβιτς ανέλαβε, επέτρεψε να δοθούν τα στοιχεία αυτά και διοργανώθηκε και μια συνάντηση με συμμετοχή μη κυβερνητικών οργανώσεων για το μέλλον του διαμεσολαβητή με τη νέα εντολή του που δέχτηκε σαφώς ότι ο χειρισμός θα μπορούσε, ε, αυτό το είπε ο Επίτροπος, είπε ότι θα μπορούσε ο χειρισμός να ήταν καλύτερος. Θέλω να το σημειώσω αυτό θετικά, παρά τη σοβαρότητα της κακοδιοίκησης κατά τη θητεία του προκατόχου του ε, τωρινού Επιτρόπου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ ο κύριο Λεγκρή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά ένα λεπτό, όχι παραπάνω. Παρακαλώ έχετε το λόγο, αλλά το πολύ ένα λεπτό. Εκτός μικροφώνου. Θα είμαι ιδιαίτερα σύντομος ε, για να απαντήσω στο σύνολο αυτών των ερωτήσεων, κάτι που είναι δύσκολο. Χαίρομαι που η υπόθεση αυτή εξετάζεται αμέσως μετά τη συζήτηση που έγινε σχετικά με το γενικότερο πλαίσιο, δηλαδή στο πλαίσιο της έκθεσης και που αφορά θέματα που, όπως η κουλτούρα της υπηρεσίας και το θέμα των νομικών απαιτήσεων και τη δυσκολία που ενδεχομένως να υπάρχει το να βρεθούμε στο σταυροδρόμι των επιμέρους συμφερόντων που προβλέπονται και προστατεύονται από τον οργανισμό 1049. Η περίπτωση αυτή δεν ε, αντικατοπτρίζει τα πράγματα γενικά. Κατα... Ε, τονίζουμε τις προσπάθειες που καταβάλει η Κομισιόν σε ζητήματα διαφάνειας, όπως ε, η ενημέρωση, το, το μητρό των ε, lobbying και βλέπουμε λοιπόν με ποιο τρόπο όλα αυτά εξετάζονται στο πλαίσιο μιας ε, δράσης που προωθεί τη διαφάνεια και που ανικατοπτρίζει την μόνιμη και συνεχή συνεργασία της Κομισιόν και εγώ που διευθύνω την υπηρεσία που διαχειρίζεται τα θέματα διαφάνειας αντικατοπτρίζουν και τις προσπάθειες που καταβάλουν οι συνεργάτες μου για να εκμεταλλευτούμε τον δυνατήριο που μας δίνει ο κανονισμός στα ζητήματα διαφάνειας όλων των εμπλεκομένων. Στη συγκεκριμένη περίπτωση και δεν θα έχω τον χρόνο να ζητήσω από τον συνεργάτη μου που είναι παίων επί του θέματος που ασχολείται με το ζήτημα αλλά αντιμετωπίσαμε μια κατάσταση που ήταν απλή στην ουσία ή θα αποφασίζαμε και να θα λέγαμε ότι θα καθιστούμε όλα δημόσια και τότε και τα κοινοποιούμε, θα θέταμε την πόρση σε μια τέτοια θέση που θα τη επιτρέπαμε να κάνει μια προσφυγή και ακόμα και σήμερα τα έγγραφα αυτά δεν θα μπορούσαν να δημοσιοποιηθούν διότι θα αποτελούσαν τμήμα του φακέλου αλλά ή θα έπρεπε να χρησιμοποιήσουμε τις δυνατότητες που μας έδιναν και να καταλήγουμε σε μια ε, λύση μετά από διαπραγμάτευση. Φυσικά μπορεί να υπάρξουν διστάμενες απόψεις αναφορικά με τη διάρκεια της όλη διαδικασία και αναγνωρίζω πως υπάρχουν κάποια στοιχεία εκτίμησης, αξιολόγησης που μας οδηγούν σε διαφορετικό αποτέλεσμα. Αλλά ε, ζητήσαμε πρόσβαση στα έγγραφα και προσπαθήσαμε να πάμε προς την οδό της απόλυτης διαφάνειας και να μπορέσουμε στο τέλος να καταστήσουμε τα έγγραφα αυτά προσβάσιμα, δημόσια, διότι φυσικά εν μέρη, διότι πρέπει να προστατεύσουμε και κάποια συμφέροντα, ε, αλλά το να αξιολογούμε αν κάποια πληροφόρηση μπορεί να ε, επηρεάσει κάποια βιομηχανικά συμφέροντα είναι ένα θέμα πολύ λεπτό και σημαντικό. Θα μπορούσα να σας εξηγήσω και να σας μιλήσω για περιπτώσεις ε, συγκεκριμένες και λεπτομεριακές ε, πρόεδρος. Ε, θα έχουμε μια συζήτηση περί αυτού. Ελπίζω πως ο καθένα στην, θα δηλαδή δει στη θέση της Επιτροπή κάποια προσπάθεια προσβολής των βουλευτών και έλλειψη συνεργασίας. Κοιτάξτε, επί του θέματος μπορείτε να επανέλθετε και να μας μιλήσετε. Εμένα μου είπατε ότι θέλατε το λόγο για να πάρει την κυρία Παλιαδέλη. Ε, φυσικά είμαι έτοιμος να εξετάσω πιο λεπτομεριακά το κοινοβουλευτικό ερώτημα που ετέθη, αλλά αυτό που θα ήταν δυνατόν, εκτός μικροφώνου, μα δεν απαντήσατε στην ερώτησή μου. Η ερώτησή μου ήταν η εξή. Γιατί δόθηκε παρόμοια απάντηση σε ένα μια ερώτηση που θα έπρεπε να απαντηθεί. Αυτή εδώ δεν είναι απάντηση. Κοιτάξτε, εγώ αυτή τη στιγμή που σας ομιλώ δεν έχω τα στοιχεία της απάντησης διότι δεν γνωρίζω την ουσία του θέματος. Άρα δεν μπορώ να εκτιμήσω την απάντηση. Φυσικά θα το εξετάσω το συντομό δυνατόν και θα σας δώσω την κατάλληλη εξήγηση. Ε, υπάρχουν πολλές εκκλησίες που μπορούν να δοθούν. Πρόεδρος, ευχαριστώ για την απάντηση που δώσετε την κυρία Παλιατέλη. Να σας ευχαριστήσω κύριε Διαμαντούρο για την εξαιρετική εργασία που κάνατε ότι κάνουν τις δύο αυτές εκθέσεις σας και θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε μαζί σας. Ευχαριστούμε και για τις απαντήσεις που δώσατε στους συναντέλφου. Αυτά να κάνω μια παρατήρηση. Μπορώ να κάνω μια μικρή παρατήρηση παρακαλώ. Προς τον κύριο που μίλησε για την ειδική έκθεση, μια μικρή παρατήρηση, σύντομη. Δέχομαι τα λεγόμενά σας και εκτιμώ ιδιαίτερα αυτά τα οποία απλωθεί να πετύχει η Κομισιόν σε ό,τι αφορά αυτή τη συγκεκριμένη έκθεση. Παραμένει μυστήριο για μένα διότι η Κομισιόν τελικά αποφάσισε να ε, δημοσιεύσει τι επιστολές γιατί χρειάστηκαν 15 μήνες πέραν των προθεσμιών και των διοριών που ήταν επιβεβλημένες. Ευχαριστώ. Με τα χαράς να σας ξανασυναντήσουμε κύριε Διαμαντούρο. Να δώσω το λόγο στον κύριο Στόκουελ εξ ονόματος ε, της ε, ο οργάνωσης Names Action for Compensation in Europe πρόκειται για την ε, αναφορά 791-2008 αφορά ε, ένα αίτημα για δικασία στην κατά την Ηνωμένου Βασιλείου για εικαζόμενη δυναμή εφαρμογής της οδηγίας 73-239 σε ε, πλαίσιο της υπόθεσης Lloyds. Καλώς κύριε Στόκουελ. Ε, έχετε πέντε λεπτά. Αν σας χρειαστούν λιγότερο, ακόμα καλύτερα. Όχι, όχι παραπάνω από πέντε όμως, διότι έχουμε και άλλο ένα σημείο με της κυρίας Γκέριγκερ. Παρακαλώ. Thank you, Madam President. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, πρόκειται για αποτυχία των δικαστηρίων στη Βρετανία να αντιμετωπίσουν το κοινοτικό δίκαιο νομίζω ότι ε, είναι πιο περιορισμένη η περίληψη που κάνετε γιατί αναφέρατε στην υποτιθέμενη αποτυχία εφαρμογής της οδηγίας σε σχέση με τους Lloyds. Αυτό ισχύει για την πρώτη αναφορά που φέραμε στο Κοινοβούλιο και την οποία στεναρός και επανειλημμένος ε, υποστήριξε το Κοινοβούλιο. Αυτό που μας απασχολεί εδώ είναι η αποτυχία των Βρετανικών δικαστηρίων να συνάδουν με την συνθήκη που είναι διαφορετική η διατύπωση αυτή από αυτή που αναφέρεται στην ημερήσια διάταξη. Πρέπει να υπενθυμίσω στα μέλη, ιδιαίτερα τα νέα, κάποια από τη μακρά ιστορία του θέματος. Το, το Lloyds είναι γνωστοί αντασφαλιστές ε, μακράς ε, ε, ιστορίας. Αναφέρθηκε ε, ότι ήταν η επένδυση αυτή που πρότειναν ασφαλής ε, με απόδοση της επένδυσης ε, μέτρια και συνεχιζόμενη. Πολλοί μπήκαν στη δεκαετία του 80 χωρίς όμως να πάρουν κάποια επιταγή και κάποια στιγμή τους ζητήθηκε να καταβάλουν τεράστια ποσά για να αντισταθμίσουν τις απώλειες. Σε ορισμένες περιπτώσεις έφτασαν στο 100% του κεφαλαίου που είχαν διαθέσει και δεν μπορούσαν να φύγουν από την αγορά πριν να περάσει, πριν να υποστούν τετραετής απώλειες. Και τώρα οι Lloyds αλλάζουν τη θέση τους και λένε ότι θα ε, παραμείνουμε ε, υπόλογοι για τις απώλειες αυτές μέχρι το τέλος της ζωής μας και ακόμη και παραπέρα. Πολλοί καταστράφηκαν, πτώχευσαν, δεν εκπλήσει ότι από πολλοί ε, ζητήσαμε να μας δοθούν εξηγήσει. Στην ε, δικαστική διαδικασία από το 1999 μέχρι το 2002 πολλές δικαστικές αποφάσεις. Το δικαστήριο συνόψη το 2000 και είπε ότι ε, είναι το χρονικό καταλόγου αποτυχιών και ανεπαρκιών στην προηγούμενη δεκαετία από τους αντασφαλιστές και άλλους ε, χρηματιστές που πραγματικά δυσφήμισαν μια σημαντική αγορά. Και ε, οδήγησαν σε προβλήματα αθωαθήματα. Παρά τις καταδικαστικές αποφάσεις, τα ονόματα, οι, οι names δεν αντισταθμίστηκαν γιατί οι Lloyds ισχυρίστηκαν ότι είχαν ασυλία ε, ε, και από το Κοινοβούλιο το 1992, το Βρετανικό, κάνοντας τις λάθος παραστάσεις στο Κοινοβούλιο όπως και στη Names. Το αποτέλεσμα είναι ότι η Lloyds είναι ένα, ε, ε, ε, ένας οργανισμός που αποκομίζει κέρδη από τέτοιου είδους καταστροφές. 18 δις ευρώ ζημιών και στοιχείων πέρασαν στο Equitest που ανέλαβε τις ιστορικές ε, ζημίες. Ε, οι Lloyd συνέχισαν και οι ε, αφανισμένοι έμειναν να φροντίσουν τον εαυτό τους χωρίς καμία αποζημίωση λόγω της, των παραστάσεων που έκαναν οι Λόιτζε. Ορισμένοι μάθαμε για τις οδηγίες ε, της Ένωσης ε, το 1997 για την αγορά και ε, στείλαμε μια αναφορά στο Κοινοβούλιο. Το Κοινοβούλιο ασχολήθηκε, η Κομισιόν όμως δεν άρχισε έρευνα πριν από το 2001. Η έρευνα εντόπισε πολλές ελλείψεις στη λογιστική των Λόιτζ και παραβιάσεις της οδηγίας 73-239. άρχισε η διαδικασία επί παραβάση αλλά το 2000 το Ηνωμένο Βασίλειο πέρασε ένα νέο νόμο που αναφερόταν που ε, ε, ίσχυσε και για τους το, το Δεκέμβριο 2001 έτσι το 2003 η Κομισιόν σταμάτησε τη διαδικασία επιβαραβάση λέγοντας ότι τώρα ε, συμμορφούνται προς το κοινοτικό δίκαιο η Βρετανία. Το κοινοβούλιο αυτό προσπάθησε να πείσει την Κομισιόν να δηλώσει σαφώς ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν συμμορφώθηκε, δεν συμμορφώθηκε το πριν από το 2001 στο κοινωτικό δίκαιο. Οπότε θα υπήρχε σαφής δικαίωση και θα ήταν πολύ καλό για την Names. Το Κοινοβούλιο ε, ε, ε, ενέκρινε την ε, έκθεση του Ρόι Πέρι που ήταν τότε ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής αυτής. Μετά ακολούθησαν δύο ψηφίσματα του Κοινοβουλίου και μια δήλωση από τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου. Ήταν πολύ ασύνθεση βήμα αυτό του Κοινοβουλίου που έδειχνε την ανησυχία του για τέτοιες κανονιστικές αποτυχίες και λήψεις σε ένα κράτος μέλος και για την ε, ανησυχία του για το τεράστιο πρόβλημα και την αδικία για τους πολίτες κατά το Κοινοβούλιο. Αναμφίβολα η Βρετανική κυβέρνηση δεν μπόρεσε να συμμορφωθεί με το κοινοτικό δίκαιο, ιδιαίτερα την ε, ε, ε, οδηγία του 1973 και από το 1978 μέχρι το 2008. Το Κοινοβούλιο και η Κομισιόν κάλεσαν τη ΝΕΙΜΣ να προσφύγει για αποζημίωση στα Βρετανικά δικαστήρια. Οι ζημιές προέρχονται από την αδυναμία εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου. Ε, όταν προσφύγαμε κατά τον Λόιτζ ε, ε αναφερθήκαμε σε ε, δόλια ε, παράσταση των Λόιτζ. και Ε, από το 81 μέχρι το 96 τουλάχιστον κατά το διάστημα αυτό οι Λόιτζοι είπαν ότι είχαν ένα λογιστικό σύστημα το οποίο και παραθέτω έκανε λογικές εκτιμήσεις για τις ε, ε, ζημίες που προβλέπονταν. Αυτό ήταν λάθος. Το 2002 λοιπόν μετά το έβριμα ότι δεν είχαν το απαιτούμενο λογιστικό σύστημα η Lodge για τουλάχιστον 15 χρόνια. Ε, μηνύσαμε τη Βρετανική κυβέρνηση για τις απώλειες ε, λόγω της ε, μη εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου. Και το Κοινοβούλιο και η Κομισιόν άλλωστε μας ενεθάρρυναν προς αυτή την κίνηση. Αυτές οι διαδικασίες προχώρησαν στα Βρετανικά δικαστήρια ε, με βάση την υπόθεση ότι το κοινοτικό δίκαιο δεν είχε εφαρμοστεί. Αυτό ε, δεν ήταν θέμα, είχε γίνει δεκτό για την ε, κροματική διαδικασία. Η Βρετανική κυβέρνηση είπε όμως ότι οι names δεν είχαν δικαίωμα να μηνύσουν τη Βρετανική κυβέρνηση και εκεί είναι ένα θέμα που πρέπει να απασχολήσει κάθε χώρα στην κοινότητα και ο κάθε πολίτη. Γιατί το δικαστήριο είπε επανειλημμένως ότι κυβερνήσεις ε, θα πρέπει να είναι υπόλογες για την αποζημίωση όταν ε, υπάρχουν απώλειες λόγω μη εφαρμογής κοινωτικού δικαίου. Αυτό είναι πολύ σημαντικό πολίτες δηλαδή που χάνουν χρήματα λόγω της ε, δυναμίας εφαρμογής ε, κοινωτικού δικαίου. Αυτοί οι πολίτες ε, πρέπει να αποζημιωθούν βεβαίως, θα πρέπει να αποδείξουν τις απώλειες που υπέστησαν σε αυτή την περίπτωση. Το Βρετανικό, τα Βρετανικά δικαστήρια ε, διαπίστωσαν ότι συνέβαινε αυτό και όταν είπαν ότι τα names ήταν αθώα θύματα. Ε, τον Λόιτσε λόγω της ε, μη υπαρξής λογιστικού συστήματος. Αυτό δεν θα ε, είχε προκύψει βέβαια αν είχε εφαρμοστεί η οδηγία τη δεκαετία του 70. Υπάρχει λοιπόν από το εφετείο απόφαση που λέει ότι οι μόνοι που μπορούν να μηνύσουν μια κυβέρνηση για αποζημίωση είναι εκείνοι όπου ε, θα έπρεπε να έχουν δικαιώματα για να εφαρμόσουν την οδηγία. Αυτό δεν είναι παράλογο, γιατί φαίνεται ότι δικαιώματα πρέπει να δοθούν μόνο σε δημόσιους υπαλλήλους που δεν ε, υπέστησαν απώλειες. Ε, η οδηγία έδωσε το δικαίωμα να προσφύγουν κατά της κυβέρνησης σε οποιονδήποτε για λόγους μη εφαρμογής οδηγίας. Αυτό είναι η πρόθεση του δικαστηρίου στη, ε, το εφετείο δεν ε, αναφέρθηκε στα θέματα αυτά. Θέσαμε ερωτήματα ε, και σε σχέση με το κοινοτικό δίκαιο, το οποίο πρέπει να αναφερθεί με βάση την, το σχετικό άρθρο της συνθήκης το Υπουργείο των Λόρδων δεν ε, αρνήθηκε να εξετάσει την υπόθεση σχετικά με το κοινοτικό δίκαιο που ετέθη, χωρίς να δώσει εξηγήσει για την άρνηση αυτή. Μετά από την άρνηση αυτή από τα Βρετανικά δικαστήρια προσφύγαμε στην Κομισιόν και κάναμε αναφορά το 2008 στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τότε η Κομισιόν έκανε μια σειρά από παραδεκτά ε, και δέχθηκε ότι η Βουλή των Λόρδων είχε παραβιάσει το θέμα. Δεν εξέτασε την αντίδραση άλλων κοινοτικών δικαστηρίων, ούτε ζήτησε το, ε, την ε, απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Όμως αποφάσισαν να μην αρχίσουν διαδικασία επί παραβάση κατά του Ηνωμένου Βασιλείου λέγοντας ότι συμφώνησαν με τα βρετανικά δικαστήρια. Πάνω σε τι δεν είναι σαφέ. Η Κομισιόν λέει λοιπόν ότι τα βρετανικά δικαστήρια θα πρέπει να, είναι, να έχουν δίκιο αφού η απόφαση ήταν ότι δεν, είχαν δικαίωμα, δεν είχε δικαίωμα η Names επειδή ε, δεν ήταν διάδικη. Δεν ε, είναι έγινε εξέταση λοιπόν. Ε, συμφωνούν, ενώ πρώτα διαφωνούσαν με τα βρετανικά δικαστήρια μετά από μια, με έναν επανορισμό σε σχέση με το ποιος έχει δικαιώματα από τα Βρετανικά δικαστήρια. Ε, μπορεί το Names όμως να είχε δίκαιο με την έννοια ότι ήταν οι μόνοι που ε, έκαναν άμεση ασφάλιση σύμφωνα με την οδηγία και ίσως ε, να έχουν δικαιώματα και να είναι οι δικαιούχοι παρόλο που δεν είναι διατεθειμένοι να κάνουν τίποτα για μια τέτοια κατάφορη παραβίαση των συνθήκων. Κυρία Πρόεδρε, δεν είναι καθόλου ικανοποιητικό το γεγονός ότι δεν μπορούν οι πολίτες να ε, θέτουν θέματα κοινοτικού δικαίου ε, στη δικαιοσύνη των κρατών μελών. Δεν είναι αυτό η πρόθεση της συνθήκης. Ούτε είμαστε μόνοι που είμαστε αγανακτισμένοι, γιατί υπάρχουν και άλλες παρόμοιες αναφορές που λέγουν ότι ε, τα βερτατικά δικαστήρια δεν λαμβάνουν υπόψη το κοινοτικό δίκαιο και για περιβαλλοντικά θέματα κυρίως και δεν τα παραπέμπουν στο δικαστήριο ενώ θα έπρεπε και ε, ε, ενδεχομένως να είχε διαφορετική άποψη από την άποψη των Βρετανικών δικαστηρίων. Έτσι έχουν ε, χαθεί δισεκατομμύρια ευρώ. Όσοι δεν έχουν πεθάνει είναι δηλικιωμένοι. 80 ετών έχουν φτάσει τα θύματα είναι ε, τα θύματα παραλήψεων, αμέλειας, ε, ε, λάθος παράστασης από τους Λόιτς. Το η Βρετανική κυβέρνηση θα πρέπει να ρυθμίζει τους Λόιτς. Όμως ένιψε τα σχήρα της αποποιούμενη κάθε ευθύνη. Τα συμφέροντα στους νέους Λόιτς που τώρα δίνουν δισεκατομμύρια στερλίνες κέρδη δεν ε, αποζημίωσαν την Names. Επίσης η δικαστική διαδικασία ε, δυσχεραίνεται από την ε, συμμετοχή της κυβέρνησης που παίζει ρόλο ε, στη, στη, στη συνεχιζόμενη αδικία και λόγω της τάσης των Βρετανικών δικαστηρίων. Εμείς ζητήσαμε τη βοήθεια του Κοινοβουλίου. Δεν θέλουμε απλά λόγια συμπάθεια. Το Κοινοβούλιο επανειλημμένα ε, παραδέχθηκε το δίκαιο των ετοιμάτων μας. Αυτό που θέλουμε είναι απόφαση από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και αν δεν τεθούν τα κέρια ζητήματα ε, από τις Βρετανικές αρχές ε, και τα Βρετανικά δικαστήρια θα πρέπει το Κοινοβούλιο να το κάνει επίσης. Ε, Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να εξετάσει το θέμα προσεκτικά η Νομική Επιτροπή να δει δηλαδή το θέμα δικαίωματος ανάληψης δράσης όταν υπάρχει ε, μια εφαρμογή κοινοτικού δικαίου όταν αγνοούνται τα δικαιώματα των πολιτών για λόγους πολιτικής σκοπιμότητας ή για άλλους πολύ σκοτεινούς λόγους. Ε, ε, με στη διάθεση της Επιτροπής, κυρία Πρόεδρε, για να απαντήσω σε ερωτήσεις. Ευχαριστώ. Δώστε λόγο στην Κομισιόν και μετά στους συναδέλφους. Παρακαλώ. Καλή σας ημέρα. Χαίρομαι που σας γνωρίζω. Θα είμαι όσο γίνεται πιο σύντομο το βασικό θέμα είναι η παράληψη των ευρωτερικών δικαστηρίων να προσφύγουν στο 10. Τα κατώτερα δικαστήρια κατέληξαν στο ότι δεν υπήρξε λόγος προσφυγής στο 10. Η δε βουλή των Λόρδων, το ανώτερο τότε δικαστήριο, συμφώνησε. Παρά το ότι δεν είπαν ρητά ότι δεν υπήρχε λόγος, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ήταν ορθά τα συμπεράσματα στο οποίο κατέληξαν οπότε θα πρέπει να επαναλάβω, το 2008 προσέφηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, ο κύριος Στόγουλ και Νέιμς, έκλεισε υπόθεση το 2009. Οπότε πρέπει και εγώ να σας ξεκαθαρίσω αυτά τα οποία είπαμε. With ε, ε, Όπω τα είπε λοιπόν ο επισυλλογητή, θα πρέπει όλα να είναι διάφανα και είχαμε επομένω ε, ε, ανταλλαγή μακρά ε, επιστολών με το, και του κυρίου ε, Μακρύβη. Είχαμε, μιλήσαμε και με τον κύριο Πέρι. Οπότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρώτα-πρώτα σε σχέση με τα όσα είχαν προηγηθεί όσον αφορά τη μη εφαρμογή τη οδηγία 73 και 79. 239 είπαμε ότι είχαμε όλο αυτό το serial που ακολούθησε και τα προβλήματα επομένω με τους names. Πάρα πολύ θλιβερή και στενάχωρη υπόθεση. Είχαμε επομένω μια μακρά ανταλλαγή ε, επιστολών και απόψεων με τον κύριο Στόκουελ, με, ε, με τον βουλευτή, τον κύριο Πέρι η εσωτερική αγορά και η νομική υπηρεσία επελήφθησαν πλευράς Επιτροπής. Βασικά πάντως η νομική υπηρεσία χειρίστηκε το θέμα. Και, καταρχήν, η Βουλή των Λόρδων θα έπρεπε να δικαιολογήσει το γιατί δεν προσευχηστό ΔΕΚ Παρ' όλα αυτά, εμείς θεωρούμε ότι αυτή η προσέγγιση, αυτή η απόφαση είναι ορθή και δεν υπάρχει αμέλεια ή ενδεχόμενος δόλος στις ενέργειες των Βρετανικών Δικαστηρίων και αυτά τα είπαμε και στην απάντηση και στην ε, απάντηση της κοινοβουλευτικής ερώτησης ή επερώτησης του κυρίου Πέρη κάποιου άλλου ευρωβουλευτού ε, που φέρει τον αριθμό 22.200 ε, κάτω στο 05. Και είναι φυσικά είπαμε θλιβερή αυτή η υπόθεση, αλλά από πλευρά κοινωτικού δικαίου δεν θεωρούμε ότι εδώ χωρεί περίπτωση παραβίαση του άρθρου 234 συνθήκη ΙΟΚ και γι' αυτό τα είπαμε και όλα αυτά που είπαμε σε αυτή την μακρά ανταλλαγή απόψεων. Οπότε και γι' αυτό και αποφασίσαμε να μην προσφύγουμε κατά του Ηνωμένου Βασιλείου. Αυτά τα είπαμε στον κύριο Στόκουελ. Έκλεισε η υπόθεση στις 8 Δεκάτου του 2009. Αυτά από πλευρά μα. Φυσικά, αν θέλετε να σα πω όλε τι λεπτομέρειε. Ο κύριο Τσίτσεστερ του έχει το λόγο. Um, can I uh, start by um, expressing a form of um, non-interest but sympathy in this issue uh, because Καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά ε, το, το τι έγινε στην υπόθεση. Θυμάμαι στην δεκαετία του 70 είχα κληθεί για να ε, γίνω και εγώ ένας από τους names στη Λόιδ και ευτυχώς, ευτυχώς τότε δεν ήμουν στη να α, αποδεχθώ μια που δεν είχα αρκετά χρήματα. Και ευτυχώ, όπω σα είπα. Παρ' όλα αυτά όμω καταλαβαίνω απολύτω το, το, πρόβλημα. Αυτό το οποίο έπληξε του νέου. Ε, και ξέρετε, ε, πολλοί ψηφοφόροι μου μου έστειλαν επιστολέ και μου εξηγούν πάρα πολλά από αυτά τα φλιβερά τα οποία έλαβαν χώρα σε αυτή την υπόθεση. Για όλο αυτό το σύριαλ που κράτησε τόσο καιρό. Και φαίνονται εκπληκτικά όλα αυτά σε κάποιον ε, που δεν είναι μέσα στο χώρο. Φίλοι μου έπεσαν θύματα της υπόθεσης αυτής, ξέρετε. Με χαρά μου ακούω ότι αναφέρθηκε και το έργο του, του φίλου Ροϊπέρη, ο οποίος επετέλεσε αξιόλογο εδώ στο κοινοβούλιο. Βοήθησε και τους names προσπάθησε τέλο πάντων να αποδοθεί δικαιοσύνη. Πάντω. από ξέρω, το κοινοβούλιο έκανε ό,τι μπορούσε για τους ε, ετούμενους. Και μεγάλη μου χαρά. Όμως, διαπιστώνω ότι συνεχίζουν τον αγώνα τους. Άρα και εμείς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μην είναι ανοιχτή η, αναφορά, η υπόθεση. Είναι κάτι σαν την Equitable Life. Και εδώ επομένω θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας. Και επίσης θέλω να επιθυμίσω στον κύριο Στόγουελ ε, και στου ε, άλλου ετουμένου ότι απεριόριστη ευθύνη σημαίνει αυτό ακριβώ που λέει. Απεριόριστη ευθύνη. Αυτό θα πρέπει να καταλάβει κανείς αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη. Γι' αυτό κατέληξαν εκεί που κατέληξαν. Οι περιστάσει αλλάζουν, η συγκυρία αλλάζει, η φορολογικό καθεστώ, Αυτό ακριβώ έμπαθαν και οι Lloyds. Και άλλαξαν πολλέ μεταβλητέ στο παιχνίδι, στην εξίσωση. επομένω, είναι υποχρεωσή μας να κάνουμε ό,τι μπορούμε, τόσο ώστε να εξωθήσουμε τι αρμόδιες αρχέ να αιτιολογήσουν τι αποφάσεις τους. Άκουσα τον εκπρόσωπο τη Κομισιόν Μα είπε την Πρεσβευτική κομισιόν και συγχαρητήρια για τα όσα κάνανε. Το οποίο ήταν πάρα πολύ λίγα και ανεπαρκή για αυτή την υπόθεση. Επομένω, ε, κάποιο θα πρέπει να ζωρίσει την Κομισιόν να κάτσει για να τα ξανασκεφτεί. Τώρα, δύο σκέψεις, κύριε Πρόεδρε. Ποιο θα πληρώσει την ύφη μια από τόσα λεφτά χάθηκαν. Ποιο θα κάτσει να αποζημιώσει όλους αυτούς τους names που υπέστησαν τέτοια ζημία. Αυτό πλευράς πρακτικής. Τώρα και κάτι άλλο. Κάτι άλλο το οποίο αφορά την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων. Υπάρχει προηγούμενο. Δηλαδή να προσφεύγει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο ΔΕΚ και να εξέτασε κάποιες υπόθεσεις. Για παράληψη που είναι υπόλογη κομισιόν ή κάποιο κράτος μέλος. Αυτό ίσως ε, είναι και ενδιαφέρον για τον κύριο Στόγκουλ και τους ε, συναυτό. Πρόεδρος, εφόσον δεν μπορώ να σας δώσω το λόγο σε κάποιον άλλο συνάδελφο, αλλά θα το συνεχίσουμε. Θα ξανασυζητηθεί αυτή η αναφορά, θα ξαναμπεί στη μέση διάταξη των συντονιστών. Να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε. Έγινε κατανοητό το πρόβλημά σας. Θεωρούμε ότι είναι θεμητά αυτά το οποίο διεκδικείται και θα πρέπει αυτό να συζητηθεί και με τους συναδέλφους της Νομικής Επιτροπής. Δεν θα δώσω σε άλλον το λόγο, διότι ήδη έχουμε καλύψει τον προηγούμενο χρόνο και τώρα η κυρία Γκέρνγκερ θα λάβει το λόγο. Και συμπαθά, συμπαθάτε λίγο σχονοσμένη κύριε Γκέρνγκερ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Το ζήτημα αυτό είναι τόσο μεγάλο δεν μπορούμε να προφύρεσουμε ένα λεπτό και να, για την παρουσίαση. Να θέσω μία ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα αναμείνουμε την απάντηση είτε σήμερα είτε αργότερα. Θα μιλήσω τώρα στην Πολωνική. Ξεκίνησε ο αγωγό φυσικού αερίου στην Βαλτική θάλασσα και στο... αυτό είναι ένα θέμα το είχαμε συζητήσει και πέρυσι στην Επιτροπή μας και είχαμε εκφράσει σημαντικέ επιφυλάξει. Ο, Όμιλος θα έπρεπε να κάνει μια εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων και αυτή η μελέτη θα έπρεπε να γίνει από ένα αυτόνομο Ινστιτούτο το οποίο θα διόριζαν όλες οι χώρες που συμμετείχαν στο σχέδιο και παράκτηση της Βαλτικής. Θα θέλω να μάθω η Κομισιόν ε, έλαβε υπόψη αυτή την ε, εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, διότι από ό,τι γνωρίζουμε αυτή τη μελέτη δεν την ανέλαβε ένα αυτόνομο, ένα ε, εξάρτητο Ινστιτούτο, αλλά ο ίδιος ο επενδυτικός όμιλος. Θα θέλαμε να μάθουμε εάν ε, οι πολίτες ε, των ε, βαλτικών χωρών θα πρέπει να κοιμούνται ήσυχοι ή θα πρέπει να ανησυχούν, διότι υπάρχουν ακόμα πάρα πολλές αμφιβολίες. Θα ήθελα μια απάντηση σχετικά με την ανεξαρτησία αυτού του Ινστιτούτου. Παρακαλώ, προς Κομισιόν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω πως ε, δεν έχουμε χρόνο για να μπούμε σε λεπτομέρειες, αλλά το θέμα είναι πολύ σημαντικό και συζητήθηκε και εδώ στο Κοινοβούλιο επανειλημμένα και σε δημόσιες ακροάσεις. Να πω πως ε, αυτό το σχέδιο είχε συμπεριληφθεί στην ε, απόφαση για τα σκαλτήρια γραμμές για τα 10 προγράμματα του 2006 μαζί με άλλα προγράμματα τώρα. Ο, ιδιώτης επενδύτης ζήτησε την υλοποίηση του προγράμματος για να μπορέσει να προχωρήσει και να το έργο θα έπρεπε να λάβει την σύμφωνη γνώμη πολλών ε, κρατών μελών ε, και χώρες από τις, από κρατών, συγγνώμη, και τις χώρες από τις οποίες ε, θα περνούσε ο αγωγός και από την αποκλειστική του ζώνη. Το Ευρωκοινοβούλιο και η Κομισιόν ενημερώθηκαν το 2007 και αυτό το οποίο συνέβη είναι πως σαφώς αναφέρεται πως, ότι με βάση την κοινοτική νομοθεσία αυτό το σχέδιο θα πρέπει να τύχει ε, εκτίμησης, ε, περιβαλλοντικής εκτίμησης επιπτώσεων σύμφωνα με την ε, οδηγία που ισχύει για την κοινοτική επικράτεια. Τώρα η Επιτροπή αυτή εξ αρχή ανέφερε πω από θεσμική σκοπιά δεν έχει να διαδραματίσει κανένα ρόλο αναφορικά με τις ανεξάρτητες αυτές μελέτες. Η ανεξαρτησία των μελετών ε, γιάται από, την, ε, από αυτή την ίδια την περιβαλλοντική εκτίμηση επιπτώσεων. Θα ήθελα να διευκρινίσω πως στη συγκεκριμένη διαδικασία χρειάζεται να λάβετε υπόψη σας πέντε περιβαλλοντικές εκτιμήσεις οι οποίε έγιναν σε εθνικό επίπεδο αλλά και την συνολική εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων που έγινε σύμφωνα με τη σύμβαση ΕΣΠΑ. Ένα παράδειγμα μόνο η γερμανική εκτίμηση περιείχε μία χίλιες ε, 600 σελίδες τεχνικών εκθέσεων, 400 σελίδες μη τεχνικού περιεχομένου, 720 σελίδες θέσεις αναφορικά με το πρόγραμμα Natura και 338 σελίδες τεχνικές πληροφορίες και 54 σελίδες που αφορούσαν την σύμβαση ΕΣΠ. Όλα αυτά λοιπόν ήταν διαθέσιμα στο κοινό. Όλα αυτά συζητήθηκαν με όλα τα κρατημέλη και τους εμπλεκομένους και η Κομισιόν αρχικά ε, ανέφερε ότι παρακολούθησε την όλη διαδικασία εκ του σύναγκες με εμπειρόγνωμονες από τα κράτη-μέλη ε, ότι έχουμε μια τέτοια συμμετοχή στην ε, Επιτροπή Περιβαλλοντικών εκτώσεων και στο τέλος της όλης διαδικασίας που πολύ σωστά αναφέρθηκε ότι ολοκληρώθηκε με την ε, χορήγηση των ε, περιβαλλοντικών αδειών. Υπήρξαν εκατοντάδες διαβουλεύσεις με τους πολίτες, ε, τους άμεσα ενδιαφερομένους. Ένα παράδειγμα να σας δώσω. Η Σουηδική περιβαλλοντική έκθεση εστάλει προς σχολιασμός στην ε, Ενεργειακή Επιτροπή, στην ε, Θαλάσσια Επιτροπή Διαχείρισης, στις ε, Σουηδικές Στρατιωτικές Αρχές, τα Σουηδική Μετρολογική Υπηρεσία, Σουηδικό Συμβούλιο Πολιτικής Χρονομιάς και ούτω καταξής. Λοιπόν, η συμμετοχή του κοινού των πολιτών ε, είχε ιδιαίτερη σημασία μέσα στο πλαίσιο της ΕΣΠΟ και οι πολίτες ε, όλων των βαλτικών χωρών ενεπλάκησαν σε αυτές τις συζητήσεις. Ε, τώρα, η Κομισιόν επανειλημμένα δήλωσε πως δεν είχε την αρμοδιότητα και δεν μπορούσε να υποκαταστήσει το θεσμικό ρόλο των κρατών μελών. Παρακολούσαμε την όλη διαδικασία, διασφαλίσαμε σε πολλές περιπτώσεις ε, πως όλα τα ζητήματα λέφθησαν υπόψη και ως παράδειγμα να αναφέρω επίσης ε, και το θέμα των ε, πυρομαχικών το οποίο ήταν πρόβλημα της εξαρχής. Κατανοείται ότι το ζήτημα της ασφάλειας του αγωγού μας απασχόλησε ιδιαίτερα και θα έπρεπε τα πυρομαχικά να ληφθούν υπόψη. Και αναλυτικές μελέτες εντόπισαν μια, μια σειρά πολεμφοδίων που θα έπρεπε να καταστραφούν μέσω διαδικασίες η οποία θα γινόταν αποδεκτή από το κοινό. Όλα αυτά λοιπόν παρακολουθούνται και ελέγχονται από υπεύθυνε ε, κυβερνητικές αρχές στα κράτη-μέλη. Μπορείτε λοιπόν να σκεφτείτε πώς η Κομισιόν για μία ανάρκη θα μπορούσε να παρέμβει και να πει αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να την ε, εξουδετερώσετε. Επίσης να πω ότι σε πολλές περιπτώσεις συζητήσεις με το κοινό και εδώ να λάβετε κατά νου ότι όλες αυτές διήρκεσαν πάνω από τρία χρόνια επανειλημμένα ακολουθήσαν μια διαδικασία βήμα προς βήμα. Το παράδειγμα της Γερμανίας παραδείγματος χάρη. Υπήρξε μια προσφυγή από δύο μη κυβερνητικέ οργανώσεις ε, στην απόφαση. Μία ήταν το WWF και ε, μετά από συζητήσεις που έγιναν με τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις ε, λήφθησαν αποφάσει και να ληφθούν περαιτέρω μέτρα και έτσι αποσύρθηκαν οι προσφυγές. τώρα, τα, οι άδειε χορηγήθηκαν μετά από όλη αυτή τη μακρά διαδικασία. Εκατοντάδες χιλιάδες σελίδων, μάλλον δεκάδες χιλιάδες σελίδων ε, τυπώθηκαν και η Κομισιόν εκτιμά πως ε, δεν χρειαζόταν να γίνει μια ιδιαίτερη μελέτη από πλευράς Κομισιόν που δεν έχει ούτε την αρμοδιότητα αλλά ούτε και την ε, δυνατότητα, την εξουσία να υποκαταστήσει τα κράτη-μέλη. Μπορούμε να σας αναφέρουμε κάθε λεπτομέρεια για τα όσα συνέβησαν. Όλες οι πληροφορίες αυτές είναι γνωστές και διαθέσιμες και Επίσης μπορούμε να σας ε, πούμε και το τι συνέβη, τις και κλπ. διότι πρόκειται για ε, δεκάδες χιλιάδες ε, σελίδων που γράφησαν περί του θέματος αυτού. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ. Πρέπει να διακόψω εδώ. Η Πρόεδρος ευχαριστεί τους διερμηνείς και οι διερμηνείς ευχαριστούν την Πρόεδρο. Δυστυχώς πρέπει να σταματήσω, κυρία Διόριγκερ, θα προτείνω να το θέσουμε σε μια προσοχή με διάταξη, αλλά εάν ε, μπορείτε να αποστείλετε στην γραμματεία τα έγγραφα στα οποία αναφέρεστε, τα οποία δεν έχουμε υπόψη μας, ε, σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Ε, σας ευχαριστώ όλους και διακόπτουμε στο σημείο της συνεδρίας.